So, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε τώρα εμείς με σημαντική καθυστέρηση αφού καθυστέρησα μέλη αλλά καθυστέρησα και η προσκεκλημένοι μας ειδικοί. Καλημέρα, αρχίζουμε χωρίς να είμαστε όλοι εδώ. Δημόσια ακρόαση σήμερα, προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους ε, καρκινογόνων μεταλλαξιογόνων στην εργασία. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό γιατί συνεχίζονται οι προσπάθειές μας να εντατικοποιήσουμε την προστασία στον τόπο εργασίας. Ε, είναι ε, περισσότεροι πολύ περισσότεροι θάνατοι τώρα λόγω επαγγελματικών νόσων και ε, πέρα από τα θέματα που πιάνει η Κομισιόν. Να καλωσορίσω τη Λέσλι Ράστον από το Imperial College στο Λονδίνο, τον Τόνι Μούσκον από το ETUC, τη Ρεμπέκα Σμίθ από το Business Europe, όμως είναι καθοδόν η Έλκε Σνάιντερ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Θα καθυστερήσει, οπότε αλλάξαμε λίγο τη σειρά. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στην Λέσλι Ράστον να κάνει την παρουσίασή της μετά τις τέσσερις ομιλίες. Η Μπαρίτα Ουλφσκογκ, η εισηγήτρια, θα κάνει μια σύνοψη και τέλος θα γίνει συζήτηση με ερωτήσεις. Η Λέσλι Ράστον παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή, για την πρόσκληση. Είμαι η Λέσλι Ράστον, επιδημιολόγος στατιστικολόγος στο Imperial College και ειδικεύομαι σε επαγγελματικούς και περιβαλλοντικούς ε, κινδύνους για την υγεία. Θα σας παρουσιάσω σύντομα το έργο στο οποίο συμμετείχα με άλλους μαζί, όπου εξετάσαμε το κόστος ενσωμάτωσης ή εισαγωγής ορίων επαγγελματικής έκθεσης και θα μιλήσω για τις 13, τους 13 παράγοντες που εξετάσαμε θα σας δώσω και κάποιες βασικές πληροφορίες, όχι τη μεθοδολογία βέβαια, αλλά θα σας μιλήσω για κάποιες αβεβαιότητες που ίσως πρέπει να λάβετε υπόψη όταν εξετάζετε τα δεδομένα. Ο στόχος αυτού του έργου ήταν να κάνει κοινωνικο-οικονομικές αναλύσεις ε, σε σχέση με την οδηγία 25 τα καρκινογόνα εξετάστηκαν, 13 εξετάζονται τώρα ε, από την οδηγία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο έχει κάνει μια ταξινόμηση εις ό,τι αφορά τα καρκινογόνα. Δεν εξετάζουμε το αν είναι το δεδομένο, εκεί έχουμε την κατηγορία. Έχουμε την ε, κατηγορία 1 που δείχνει ότι έχει πολύ, ε, πολλά αποδεικτικά στοιχεία το 2α η κατηγορία αυτή είναι πιθανή, δεν είναι τόσο αποδεικτικά τα στοιχεία και το 2β ε, που είναι πολλά εδώ στον κατάλογο των 25, εδώ είναι λίγα τα δεδομένα για τον άνθρωπο. Όπως είπαμε λοιπόν, εξετάζομαι τον αντίκτυπο της εισαγωγής ή μείωσης των ορίων επαγγελματικής έκθεσης και ένα θέμα είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε το κόστος και τα ωφέλη και για τη βιομηχανία. Εμείς θεωρούμε, ε, κάναμε εκτίμηση του φόρτου του επαγγελματικού καρκίνου στην Βρετανία. Πολύ σύντομα θα εξηγήσω τη γενική μεθοδολογία που αφορά στη μελέτη που κάναμε για σας. Εξετάζομαι καταρχήν προηγούμενη επαγγελματική έκθεση και σε ποιο βαθμό προκάλεσε καρκίνο τώρα. Δηλαδή τι ποσοστό καρκίνων προκαλούνται από προηγούμενες εκθέσεις. Και μετά αναπτύσσουμε μεθοδολογίες για να ε, προβλέψουμε στο μέλλον, όλο και περισσότερο στο μέλλον, πόσα ακρούσματα θα είχαμε κάτω από συγκεκριμένα σενάρια. Και συγκρίνουμε το να μην κάνουμε τίποτα με διάφορες παρεμβάσεις. Στην ε, μελέτη εξετάσαμε ε, Στη Βρετανική μελέτη είδαμε τη βελτίωση της συμμόρφωσης ε, σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας κλπ. Ε, είναι πιο περίπλοκες οι επεμβάσεις της, μετα... της Βρετανικής μελέτης. Η μελέτη αυτή σας επιτρέπει να δείτε και ε, κενά στα δεδομένα, στα στοιχεία. Το έγγραφο που ετοιμάσαμε θα σας δείξει ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις ό,τι αφορά τα στοιχεία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ιδέες για την έρευνα και δυνατότητες επεμβάσεων για τη μείωση των κινδύνων. Οι μελέτες αυτές σας δείχνουν πολλά δεδομένα. Αν πρόκειται να λάβετε απόφαση πρέπει να δείτε πολλά στοιχεία. Και εξαρτάται, τι σας ενδιαφέρει πιο πολύ. Αν σας ενδιαφέρει να μειώσετε την επαγγελματική έκθεση που όντως προκαλεί τους περισσότερους καρκίνους, τότε πρέπει να δείτε το καταλογισμό του κλάσματος. Σας ενδιαφέρουν οι θάνατοι. Πόσοι θάνατοι οφείλονται σε αυτούς τους καρκίνους λόγω των επαγγελματικών καρκινογόνων. Αν δεν σας ενδιαφέρουν οι θάνατοι, μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα νέα κρούσματα καρκίνου. Η, ε, η επίπτωση των καρκίνων δηλαδή. Επίσης, Μπορεί να σας ενδιαφέρει το εξή, Εάν έχω έναν επαγγελματικό καρκίνο, τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους θανάτους. Σημαίνει ότι θα πεθάνω νωρίς. Πόσα χρόνια ζωής θα χάσω ή αν επιβιώσω τι σημαίνει αυτό σε σχέση με κάποια αναπηρία ενδεχομένως που θα πρέπει να αποδεχτώ. Υπάρχουν πολλά μέτρα. Στην ε, μελέτη της έντοσης εξετάσαμε και τα θέματα αυτά και το κόστος τους. Θα σας δείξω λοιπόν εν συντομία τι ε, είδαμε στη Βρετανική μελέτη. Εδώ έχουμε τον καταλαγισμό των κλασμάτων, τα ποσοστά, ε, εδώ είναι οι στήλες Βλέπετε τους διάφορους καρκίνους, στο μεσοθυλίωμα περίπου 90% φτάνει και οφείλεται σε επαγγελματικούς ε, κινδύνους προκειμένου λόγω αμοιάντου μάλλον και είναι 5,3% όλων των καρκίνων γενικά οπότε εδώ έχουμε 8.000 θανάτους 13,5 80.000 ε, ε, θανάτους ή 13,5 είναι αποδεδειγμένα επαγγελματικοί. Ε, εδώ μια άλλη ε, διαφάνεια δείχνει τα βασικά καρκινογόνα, ο αμίαντος, εδώ είδαμε τις ε, βάρδιες, το διοξίδιο της πυρητίας είναι ένα που το εξετάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώστε εδώ ότι όπως και στη μελέτη της Ένωσης, ο κατασκευαστικός τομέας επιβαρύνεται πάρα πολύ με 56% μια ιδέα πώς εσείς μπορείτε να το δείτε το θέμα ως υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων. Εδώ είναι μια κατανομή στην αριστερή στήλη. Βλέπετε διαφορετικούς καρκίνους όταν δείτε το κλάσμα που καταλογίζουμε σε σχέση σε σύγκριση με ε, την, την καταχώρηση των νέων καρκίνων, ε, έτη ε, χαμένα κλπ. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε πολλούς καρκίνους του ε, πνεύμονα που είναι μοιραίος ως των θανατηφόρος. Αν σας ενδιαφέρει η μακρά επιβίωση ή σχεδόν θανατηφόροι καρκίνοι, τότε ε, πάνω στον κατάλογο θα βάλουμε τους καρκίνους του δέρματος, που δεν είναι μελανόματα, και τους καρκίνους του μαστού που έχει καλή πρόγνωση. Και βλέπουμε 10-15 χρόνια ε, έτη απολεσθέντα. Το SICAN Project, λοιπόν, δεν θυμάμαι γιατί επιλέξαμε αυτό το ακρόνιμο. Δεν θυμάμαι και τι σημαίνει πια. Πέρασε καιρός. Εξετάζαμε πάντως 25 καρκινογόνους παράγοντες. 25, 26, 27, δεν θυμάμαι πόσο αρχίσαμε. Α, όχι, συγγνώμη, σε 27 κράτη-μέλη είχαμε πολλά προβλήματα με τα δεδομένα. Δεν είδαμε μόνο τη δουλειά που κάναμε για την Βρετανική μελέτη, αλλά είδαμε και κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο. Συζητήσαμε με εμπλεκομένους, είδαμε τα επίπεδα έκθεσης ε, και πώς αντιμετωπίζονται στις διάφορες διαργασίες. Οι ουσίες, ε, ελπίζω να το διαβάσετε αυτό, αριστερά τα έχω καταγράψει με τη σειρά της καταξινόμησης του ΙΑΡΚ. Υπάρχουν 7 καταξινομήσεις 1 που είναι σίγουρα καρκινογόνα, υπάρχουν 2, α που είναι πιθανές και 5 που είναι δυνατές, λίγα δεδομένα για τον άνθρωπο τα δύο, στα 2B. Προκαλούν διαφόρους καρκίνους και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να το θυμάστε. Ο πνεύμονας εμφανίζεται πολύ στην Βρετανική μελέτη πάνω από 20 καρκινογόνα για τον πνεύμονα. Πολλά επαγγελματικά καρκινογόνα πλήττουν τον ε, πνεύμονα. Ή τιμές έκθεσης, ε, επαγγελματικής έκθεσης. Κάποιες έχουν αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αλλού σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τιμές που έχουν θεσπίσει κάποια κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν πολλοί όμως που είναι εκτεθειμένοι τώρα πάνω από αυτές τις τιμές. Αν δούμε για παράδειγμα την υδραζίνη κάτω, οι μικρότερες τιμές ε, δείχνουν ότι το 75% των εργαζομένων έχουν έκθεση σε, σε αυτή τη δήμη. Ή αν δούμε ε, την βουταδίνη, βουταδιένη, βλέπουμε 46% ε, για τις 25 ουσίες. Αλλά εδώ έχουμε και την ε, σημαντική περίοδο έκθεσης ε, κάτω από την οποία αν εκτεθούν μπορούν να πάθουν, θα πάθουν καρκίνο. Είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να δούμε και τον χρόνο που χρειάζεται για να εμφανιστεί ο καρκίνος. Πολλές φορές οι καρκίνοι εμφανίζονται μετά τη συνταξιοδότηση. Δεν θα τους δούμε όταν δουλεύουν. Θα τους δούμε μετά την, το τέλος της απασχόλησης. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί πρόβλημα ανείχνευσης, εντοπισμού του καρκίνου. αριθμού των εργαζομένων, αυτό είναι για τον τωρινό φόρτο του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι είναι σημαντικός για, τις, για τους 25 παράγοντες. Αυτή είναι η, ε, τα αρχικά δεδομένα. Αν δεν κάνουμε τίποτα απολύτως, πόσους καρκίνους θα έχουμε τώρα και στο μέλλον. Το τώρα είναι το 2010 βέβαια. Και βλέπετε ότι ε, τα βάζουν σε σειρά προτεραιότητας η σπνεύσιμη κρυσταλλική πυρητεία περίπου 7.500 καρκίνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και αν δεν γίνει τίποτε και διατηρηθεί το παρόν καθεστώς και δεν αλλάξει το όριο έκθεσης, θα είναι περίπου 450.000 τα επόμενα 60 χρόνια. Οι θάνατοι παραμένουν οι ίδιοι για την ε, πυρητεία, για την εκαρκίνωση του πνεύμονα που είναι ε, δυστυχώς σχεδόν πάντα θανατηφόρος. Και υπάρχουν σημαντικά νούμερα για τις προβλέψεις μας παντού και για τη σκόνη των σκληρών ξύλων και το χρώμιο 6. Αν δεν κάνουμε τίποτα θα χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εδώ είναι το κόστος ε, όφελος για την υγεία σε σχέση με το κόστος συμμόρφωσης. Έχουμε τα, ε, 7 ουσίες. Η δεύτερη στήλη σας δίνει ένα τομέα που έπρεπε να εξετάσουμε, τον επιλέξαμε. Βλέπετε ε, πόσα ε, κρούσματα αποφεύχθηκαν. Αν πάρουμε ας πούμε την πυρητεία 0,5 το κατώτερο επίπεδο αποφεύγουμε περίπου 110.000 θανάτους ε, αλλάζοντας το όριο. Είναι το 25% των εργαζομένων αυτοί που έχουν έκθεση στην πυρητεία. Οπότε θα είναι περισσότερα τα νούμερα έκθεσης στο κατώτερο επίπεδο που ε, ενέχουν κινδύνους επίσης, αν και μικρούς κινδύνους. Ε, η ευθεία γραμμή σημαίνει δεν υπάρχει έκθεση, δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά πάντα σε, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος σε οποιαδήποτε έκθεση. Ε, αν δούμε το συνολικό όφελος για την υγεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάποια αέρια όρια, ιδιαίτερα για το χρώμιο 6 και την ε, πυρητεία, αλλά υπάρχουν και σημαντικά κόστη συμμόρφωσης. Το, ο λόγος δηλαδή όφελος προς κόστος ε, είναι σημαντικός για την πυρητεία, το χρώμιο και τη, ε, τη σκληρών ξύλων. Στις άλλες ουσίες είτε έδειξε ότι δεν υπάρχει τιμή που να αφορά την επίπτωση στην υγεία από, την, ε, από τα όρια ε, ή φαίνεται ότι θα υπάρχει κόστος συμμόρφωσης. Οι άλλοι έξι παράγοντες, πιθανά καρκινογόνα, εκεί δεν υπάρχει όφελος για την υγεία. Ποια είναι η αβεβαιότητα εδώ. Παρουσιάζεται στο έγγραφο για τον αντίκτυπο, αλλά καμιά φορά πρέπει να είμαστε λίγο τολμηροί με τις υποθέσεις μας, με βάση αυτά που έχουμε. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το χρονικό διάστημα πριν εμφανιστεί καρκίνος, πριν από πόσο διάστημα χρειάζεται, πόση έκθεση χρειάζεται, για πόσο διάστημα. Κάναμε κάποιες υποθέσεις εδώ. Αν χρησιμοποιήσαμε δημοσιευμένα στοιχεία για αξιολογήσεις επικινδυνότητας, ε, δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι, μπορεί τα αποτελέσματα αυτών των μελετών να μην αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό που εξετάζομαι. Υπάρχουν πολλές ανακρίβειες και αβεβαιότητες σε όλα τα δεδομένα τα πληθυσμιακά και στις καταχωρήσεις των καρκίνων και υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα ε, για τους επαγγελματικούς κίνδυνου. Πάντως τα δυνατά σημεία της μελέτης είναι ότι σας δίνουν πολλά αντικειμενικά μέτρα μέτρησης, μεθόδους μέτρησης. Και εσείς, οι πολιτικοί που θα πάρετε τις αποφάσεις, θα δείτε τι σας ενδιαφέρει. Ε, ενημερώνονται και οι ε, κλάδοι της βιομηχανίας, ε, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Θέλω να πω ότι ευαισθητοποιούν γενικότερα για το θέμα των επαγγελματικών κινδύνων. η ευαισθητοποίηση αυξήθηκε πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η υγεία δηλαδή απασχολεί πολύ περισσότερο τους εργαζομένους. Ένα άλλο σημαντικό που αναφέρεται και στο κείμενο για τον αντίκτυπο είναι η, ότι η μείωση των καρκινογόνων επηρεάζει και άλλα προβλήματα ε, και αν μειώσετε την πυρητεία μειώνεται η ε, περιορισμένη λειτουργία των πνευμόνων και γενικότερα οι πνευμονοπάθειες ε, μειώνονται. Τώρα, ορισμένα πράγματα που θα ήθελα να πω σε προσωπική βάση. Ε, για τις παραλήψεις του κειμένου για τον αντίκτυπο. Ε, γίνονται συζητήσεις σχετικά με το αν πετύχαμε το στόχο και αν θα έπρεπε να θεσπιστούν συστήματα παρακολούθησης για τις επαγγελματικές νόσους. Είναι δύσκολο αυτό. Ένας ε, ογκολόγος ε, ε, του αναπνευστικού δεν θα μπορεί να πει πού ακριβώς οφείλεται ο καρκίνος. Δηλαδή δύσκολα θα αποφανθεί και θα πει ότι ναι, φταίει η πυρητεία. Όχι πάντα τουλάχιστον. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καρκίνους, ίσως το πνεύμονας δεν είναι καλό παράδειγμα, αλλά οι περισσότεροι καρκίνοι αυτοί είναι δύσκολοι. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να προσδιοριστεί. Αυτό που συστήνουμε εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι να παρακολουθείτε η έκθεση στο μέλλον. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι μας ζήτησαν να δούμε δυσανάλογα μειονεκτήματα στα κράτη-μέλη, στη βιομηχανία και κλπ. Δεν βλέπω κάποια δυσανάλογα μειονεκτήματα στο ε, ε, ε, εργατικό δυναμικό που αναφέρεται στο ε, έγγραφο για τον αντίκτυπο. Ίσως η Κομισιόν θα πρέπει να σκεφτεί μήπως... Α, δεν αναφέρεται πολύ το εργατικό δυναμικό και θα πρέπει να δούμε μήπως υπάρχουν δυσανάλογα μειονεκτήματα για το εργατικό δυναμικό. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τη δεύτερη ειδήμονα, Έλκε Σνάιντερ, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Υγείας και Ασφάλειας ε, στον τόπο εργασίας. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε και έχετε τον λόγο. Ε, ε η δυνατόν 10 λεπτά παρακαλώ. Microphone, I would first like to thank Mr. Handel and Mrs. Ευχαριστώ τον κύριο Χέντελ και την κυρία Ούλσκοφ που καλέσατε το φορέα μας να κάνει μια ομιλία σε αυτή την ακρόαση. Συγγνώμη που άρχισα, Ναι, μεν είμαι ε, ειδήμων σε τεχνικά θέματα, αλλά δυστυχώς έκανα λάθος ε, στο σημείο που περίμενα να με συνοδεύσουν να μπω στο Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα να σας δείξω μερικά βασικά στοιχεία που υποθέτω αναφέρθηκαν και από την προηγούμενη ομιλήτρια και μετά να σας δώσω παραδείγματα από τα πορίσματα των ε, μελετών που έχουμε κάνει ως φορέας και να αναφέρω και τις δραστηριότητες μας για τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά στοιχεία. Ο καρκίνος είναι ο δεύτερος κύριος ε, λόγος θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτος είναι τα καρδιοαγγειακά. Ένα από τους τέσσερις θανάτους ε, στην Ένωση οφείλεται σε καρκίνο. Και για τα άτομα κάτω των 65 είναι ένας από τους τρεις. Λοιπόν, πολύ σημαντικός λόγος θανάτου. 4 με 8% των ε, ε, επαγγελματικών καρκίνων θεωρείται ότι προκαλούνται από καρκινογόνες ουσίες στον τόπο εργασίας, αλλά δεν είναι βέβαια οι ίδιες ουσίες. Για τον αμίαντο θα ήταν 85% το ποσοστό και για κάποιους καρκίνους που προκαλούνται από σκόνες ξύλου, στη Γαλλία έχουμε μία εκτίμηση ότι είναι περίπου 50% για 50% δηλαδή των καρκίνων από τη σκόνη ξύλου πρόκειται για έκθεση για επαγγελματικούς λόγους. Το κόστος των επαγγελματικών καρκίνων εκτιμάται σε περίπου 334 δις ευρώ, αλλά είναι μια ευρή εκτίμηση. Είχαμε μια έκθεση που παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση της Ολλανδικής Προεδρίας τον περασμένο Μάιο, όπου παρουσιάστηκαν αυτά τα στοιχεία. Είναι εκτιμήσεις βέβαια, αλλά μας βοηθάνε να καταλάβουμε. Κάθε χρόνο έχουμε 102.500 θανάτους από επαγγελματικού καρκίνους στην Ευρώπη των 28 και αυτό εκτίμηση σε μια έκθεση από τον προηγούμενο διευθυντή μας, το Γιου Κατάκαλα. Και υπάρχει ένα άρθρο που έχουμε δημοσιεύσει που εξηγεί πώς καταλήγουμε σε αυτές τις εκτιμήσεις. οι επαγγελματικές καρκινογόνες ουσίες ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε πολλές παράλληλα. Οπότε υπάρχει η κενή επίπτωση διαφόρων. Για την οδηγία εξετάζουμε μία-μία τις ουσίες, αλλά ο εργαζόμενος μπορεί να εκτίθεται σε διάφορες. Να μερικά παραδείγματα. Δύο παραδοσιακών ε, εργασιών ε, σε εργοστάσια, αλλά και ορισμένοι που εργάζονται σε παροχή υπηρεσιών, για παράδειγμα παραγωγή υποδημάτων ή κομμωτές. Είναι σημαντικό λοιπόν να το ξέρουμε αυτό όταν εξετάζουμε τις επιπτώσεις. Όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι οι ουσίες που έχουν διαφόρων τύπων επιπτώσεις πρέπει να συνυπολογίζονται. Έχετε εδώ μερικά παραδείγματα από το κατάλογο ουσιών, ε, πυρητεία, ακριλαμίδι, ενώσεις χρωμίου. Έχουν και άλλα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, γίνεται κανείς πιο ευαίσθητος σε διάφορες ουσίες, ε, ε, επίσης μπορεί να γίνουν πιο ευαίσθητοι σε διάφορες άλλες ουσίες, να μειωθεί η λειτουργία των πνευμόνων τους. Οπότε αν αποφευχθεί η έκθεση θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Η ευαισθητοποίηση για παράδειγμα είναι κανείς πιο ευερέθιστος σε ορισμένες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι Ορισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να είναι ασθενείς συχνότερα και αυτό έχει υψηλό κόστος. Άρα συνολικά οι επιπτώσεις ε, ίσως να υποτιμούνται, διότι αν αποφευχθεί η έκθεση αυτή δεν θα αποφευχθούν μόνο οι καρκίνοι, αλλά και άλλες παρενέργειες. Τώρα, μερικά πορίσματα μιας μελέτης που κάναμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικά χρόνια, Δημοσιεύσαμε μια έκθεση, μπορείτε να τη δείτε στο site μας. Κάναμε μια μελέτη, μια έρευνα στα κράτη-μέλη. Ρωτήσαμε τα κράτη-μέλη να μας ενημερώσουν για τις μεθόδους πούμε, που έχουν τα κράτη-μέλη για να ορίζουν τα ανώτατα όρια έκθεσης σε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες. Και τι είδαμε ότι ποικίλουν κατά πολύ οι ουσίες και οι ε, οριακές τιμές έκθεσης. Ε, σε ορισμένες ε, περιπτώσεις, αντί να έχουμε τρεις ή τέσσερις τιμές, είχαμε μέχρι και 50 έως 60. Πολύ διαφορετική λοιπόν η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Πολλά κράτη-μέλη μας είπαν ότι έχουν απλώς μεταφέρει τα όρια από άλλες χώρες άρα βασίζονται σε πόρους άλλων για να καθορίζονται τα όρια, αλλά οι πόροι γενικά αυτοί είναι περιορισμένοι. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ακόμη πιο σαφές, είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές σε ανοσιακό επίπεδο, κοινή στόχη πρόληψης. Φυσικά, τα όρια αυτά πρέπει να επιτευχθούν μέσω μέτρων πρόληψης, καλύτερος εξαρισμός, για παράδειγμα, κλειστά συστήματα και άλλα. Δημοσίευσαμε και μια άλλη έκθεση πριν από δύο χρόνια για τα συστήματα επιτήρησης. Το ανέφερε και αυτό η προηγούμενη ομιλήτρια όπου είπε ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία και επίσης τόνισε ότι τα περισσότερα στοιχεία έχουν να κάνουν με ε, εργαζόμενους ε, στον βιομηχανικό κλάδο και όχι ε, με εργαζόμενους στις υπηρεσίες που είναι 70% και πολύ ευάλωτοι εργαζόμενοι, ομάδες ευάλωτων εργαζομένων που εκτίθενται σε καρκινογόνες ουσίες δεν εκτιμώνται σωστά. Για παράδειγμα, οι νέοι εργαζόμενοι, αυτοί που κάνουν συντήρηση κτηρίων ή άλλων εγκαταστάσεων, Υπάρχει μια μελέτη στη Γαλλία που γίνεται από ιατρούς που ειδικεύονται στις επαγγελματικές νόσους. Προσπαθούν να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα της έκθεσης ορισμένες καρκινογόνες ουσίες και διαπίστωσαν ότι αυτοί που εκτίθεται περισσότερο είναι αυτοί που ασχολούνται με εργασίες συντήρησης. Εκεί περίπου 40% εκτίθεται και οι νέοι εργαζόμενοι επίσης εκτίθεται πολύ περισσότερο από ότι οι μεγαλύτερες ηλικίε. Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους εργάζονται υπό συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες γιατί αλλάζουν τόπο εργασίας και επίσης μεταξύ αυτών των νέων υπάρχουν και πολλοί μαθητευόμενοι, δηλαδή πολλοί νέοι μεταξύ 15 και 18 ετών. Και γενικά εκπαιδευόμενοι. Και για την εργασία τους υπάρχει πολύ μικρός βαθμός ελέγχου. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε στην έκθεση είναι ότι είναι περιορισμένες ε, οι μέθοδοι για να επανέλθουν στην εργασία οι καρκινοπαθείς. Ε, μελετάμε αυτή τη στιγμή ένα έγγραφο που θα καταλήξει σε συστάσεις για αυτό το θέμα. Επίσης, ε, χρειάζονται λύσεις στον τόπο εργασίας. Θα επανέλθω. Ένα παράδειγμα μία από τις ουσίες που είναι στην ε, έκθεση, το διοξείδιο του πυρητίου, παίζει μεγάλο ρόλο. Κάποιες μελέτες ε, καταδεικνύουν, μια φιλανδική για παράδειγμα, που μελετάει τις τάσεις από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και την παρούσα, διαπίστωσε η μελέτη ότι μειώνεται η έκθεση αλλά αυτή η μείωση μοιάζει να σταματάει και εκτίθενται όλο και περισσότεροι. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τον αριθμό των ατόμων που εκτίθενται για το διοξείδιο του πυρητίου. Ε, πολλοί μπορεί να εκτίθενται παρόλα αυτά. Τώρα, τι προβλέπουμε για το μέλλον. Έχουμε παραγγείλει είμαστε καλύτερα στη φάση παραγγελίας μιας μελέτης επιπτώσεων για την έκθεση στους ε, παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο. Το πρώτο βήμα είναι να δούμε εάν μπορεί να γίνει μια τέτοια μελέτη. Είναι μελέτη ε, εφικτότητας θα για να προτείνουμε ένα κατάλογο των κινδύνων καρκίνου και να δούμε αν μπορεί να γίνει μια πιλωτική, ε, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για αυτή τη μελέτη. Να δούμε αν θα γίνει του αναδόχου. Θα τελειώσουμε ελπίζω για αυτή τη μελέτη το δεκαοχτώ. ή όλα τα κράτη-μέλη είμαστε σε φάση επιλογής ε, του αναδόχου. Θα ε, τελειώσουμε, ελπίζει, αυτή η μελέτη το 18. Οι μέθοδοι θα βασίζονται σε έρευνες που έχουν γίνει στην Αυστραλία. Είμαστε σε στενή επαφή με τους ε, ειδικού που έκαναν αυτή την ε, μελέτη στην Αυστραλία. Επίσης μια άλλη δραστηριότητα είναι η εκστρατεία μας για ε, υγιείς τόπους εργασίας, όπου θα εστιάσουμε σε κινδύνους από επικίνδυνες ουσίες, άρα εν μέρη και για καρκινογόνες ουσίες. Είναι μια εκστρατεία καλών πρακτικών Δηλαδή να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών για νέα μέσα και μεθόδους και για να αυξηθεί και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, ιδιαίτερα για τις καρκινογόνες. Η επικοινωνία σε όλη την φάση των αλυσίδων ε, παραγωγής και διανομής μας ενδιαφέρει. Σχετίζεται λοιπόν και με το REACH. Υπάρχουν κάποιοι νέοι κίνδυνοι. Κάναμε μια μελέτη το 2003 Έκτοτε έχουν υπάρξει πολλές νέες εξελίξεις, υπάρχουν τα νάνο υλικά, η έκθεση σε αυτά κτλ. Και πρέπει και εδώ να δούμε θέματα ε, ευάλωτων ομάδων και θέματα φύλου. Θα δούμε δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους για τις ε, ευάλωτες ομάδες και τις γυναίκες. Υποστηρίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως EU όσα και το νοδικό χάρτη για τις κακινογόνες ουσίες. Έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους την, ε, της υπηρεσίας της Ολλανδίας και της Αυστρίας ένα σύμφωνο δραστηριοτήτων για να βελτιωθεί η πρόληψη των επαγγελματικών καρκινογόνων. Έχουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 17 και το 18 και ίσως και το 19. Μία από τις πρώτες δραστηριότητές μας θα είναι να υπάρχει ένας οδηγός που θα δημοσιευθεί τέλη Οκτωβρίου από την Επιτροπή των ε, Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας για τους κινδύνους έκθεσης στην Πυρητία. Ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά επίσης έχουμε δεσμευθεί να υπάρχει ετησίως ε, μια εκδήλωση για συγκεκριμένες ουσίες ή συγκεκριμένους κινδύνους και να ενημερώσουμε και για όλες τις ενέργειες που θα γίνονται σε κάθε φάση μέσω του οδικού χάρτη. Καταλήγοντας, να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς άλλη καθυστέρηση προχωρούμε στον επόμενο μιλητή Τόνι Μούσου, ερευνητή από το Ινστιτούτο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο Τόνι Μούσου από το Ερευνητικό Κέντρο της ETUC που συμπεριλαμβάνει όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Λοιπόν, θα αρχίσω και περιμένω να διευθετήσω τις διαφάνειες πρώτα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εάν δούμε τον αριθμό θανάτων με βάση το, την έκθεση, την επαγγελματική έκθεση βλέπουμε ότι ένα 53% ε, μπορούν να πληγούν από την ε, επαγγελματική αυτή έκθεση και μπορώ να σας πω ότι ο αριθμός που μας έδωσε η Λέσλι Ράστον για την επαγγελματική έκθεση προκαλεί το 5 8% ε, των θανάτων και των καρκίνων. Όλα αυτά ενέχουν ένα πολύ υψηλό κόστος για την κοινωνία, για τους εργαζόμενους, για την οικογένεια, για τους εργοδότες και για την κοινωνία. Και μία πρόσφατη μελέτη από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Υγείας στην Ολλανδία μας ε, δίνει ένα συνολικό κόστος 334 δισεκατομμύρια ετησίως για την Ευρώπη των 28 κρατών τεράστιο λοιπόν το κόστος. Γι' αυτό τα συνδικάτα έχουν κινήσει μία εκστρατεία για να σταματήσει ο καρκίνος στον χώρο εργασίας. Και ένας από τους λόγους είναι το ότι όλοι αυτοί οι καρκίνοι μπορούν να προληφθούν εάν οι εργαζόμενοι δεν εκτεθούν ή εκτίθενται λιγότερο σε επικίνδυνες ουσίες. Ένα από τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υγεία για να ελαχιστοποιήσουμε τα επίπεδα αυτά έκθεσης είναι ακριβώς οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης γι' αυτό και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικαιροποιήσει τα στοιχεία των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών και να ορίσει 50 ουσίες για τις οποίες θα υπάρχουν δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης, ξεκινώντας από φέτος. Και 50 ουσίες κατά προτεραιότητα μέχρι το 2020. Βλέπετε εδώ τα αιτήματα των συνδικάτων. Η Επιτροπή πρότεινε ε, καταρχήν 13 ε, καρκινογόνες ουσίες με δεσμευτικές οριακές τιμές και εμείς θα θέλαμε να υπάρχουν πιο ε, περιοριστικές οριακές τιμές, ιδιαίτερα για τις ε, κρυσταλλικές, για το κρυσταλλικό πυρίτιο που εισπνέει κανείς για, την, ε, για τις ενώσεις χρωμίου, για την βουταδιένη και για τις πυρήμαχες κεραμικές ίνες, καθώς και τη φορμαλδεΐδη. Όπως ξέρετε υπάρχουν ε, χαμηλότερες οριακές τιμές, γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Εάν κάτι είναι εφικτό σε μία χώρα, είναι εφικτό και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε τι γίνεται με το χρώμιο 6. Έχουμε ένα εκατομμύριο εργαζόμενους που εκτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται λόγος για 25 μικρογραμμάρια ανακυβικό μέτρο, ενώ στη Γαλλία και την ε, Γερμανία, καθώς και στην Ιταλία, έχουμε ένα μικρογραμμάριο. Και ξέρουμε ότι ε, για αυτή την ουσία η Επιτροπή θα ήθελε να κάνει βήματα προς τα εμπρός. Και αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες για να έχουμε χαμηλότερες οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να έχει χαμηλότερες οριακές τιμές για τις καρκινογόνες αυτές ουσίες. Γιατί όταν συμπεριληφθούν στην οδηγία είναι δύσκολο να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε εξ αρχής να έχουμε ε, χαμηλότερες οριακές τιμές που να προστατεύουν περισσότερο τους εργαζόμενους. Η πρόταση της Επιτροπής αφορά τις αλλαγές στο παράρτημα 3, δηλαδή να προσθεθούν οριακές τιμές για ορισμένες καρκινογόνες ουσίες. Θα θέλαμε όμως εμείς με αυτή την αναθεώρηση να αλλάξουμε και ορισμένα από τα άρθρα της οδηγίας και τα συνδικάτα θα ήθελαν και το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας να επεκταθεί και σε ουσίες οι οποίες είναι ε, τοξικές για το, την αναπαραγωγή. Και θεωρούμε ότι ότι έχουμε 2 έως 3 εκατομμύρια εργαζομένους που εκτίθενται σε καρκινογόνες ουσίες και δυστυχώς η νομοθεσία είναι πολύ ήπια και αδύναμη. Δηλαδή έχουμε την οδηγία για τις εγκυμονούσες γυναίκες, όταν λοιπόν ο, εργαζόμενος, ο εργοδότης με ξέρει ότι εγκυμονεί μία εργαζόμενη, θα πρέπει να αναλάβει δράση για να μειωθεί η έκθεση αυτής της εργαζόμενης σε καρκινογόνες ουσίες. Αλλά αυτό γίνεται πολύ αργά. Δηλαδή γίνεται τρεις μήνες μετά όταν κοινοποιεί την εγκυμοσύνη και στο μεταξύ έχει εκτεθεί. Επίσης, καλυπτόμαστε από την οδηγία χημικών ουσιών και εδώ οι οριακές τιμές δεν είναι δεσμευτικές, είναι ενδεικτικές. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτές ε, τις ουσίες και στην οδηγία για τις ε, καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες για να προστατεύσουμε και την αναπαραγωγική υγεία. Γιατί ε, πολλές ε, ε εθνικές νομοθεσίες έχουν ε, συμπεριλάβει αυτές τις ουσίες ε, ανα, αναπαραγωγικής τοξικότητας, κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε γενικότερα. Υπάρχουν όμως και άλλες διατάξεις που θα θέλαμε να βελτιωθούν και αυτό αφορά και τη διαφάνεια που υπάρχει σε σχέση με την έκθεση σε κίνδυνο με βάση τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης. Το ότι έχουμε μια οριακή τιμή δεν σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης κάλυψη. Ελοχεύει πάντα κίνδυνος και αυτό που μας καλύπτει είναι η οριακή τιμή, η οποία θα πρέπει να εγγράφεται στην νομοθεσία, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με την οριακή τιμή. Επίσης, θα θέλαμε να υπάρχει ένα εποπτικό υποχρεωτικό καθεστώς της υγείας του εργαζόμενου μετά τη ε, συνταξιοδότηση. Γιατί ξέρετε ότι μεσολαβεί μεγάλο, μακρύ χρονικό διάστημα μεταξύ της έκθεσης και της εκδήλωσης του καρκίνου. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα καθεστώς εποπτείας και παρακολούθησης για να δούμε κατά πόσο αυτή η έκθεση οδηγεί σε καρκίνο. Επίσης χρειαζόμαστε περισσότερα υποχρεωτικά στοιχεία για την έκθεση, την επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες. Όταν έχουμε οριακές τιμές, χρειάζεται πολλής χρόνος για να αναθεωρηθούν. Γι' αυτό θα θέλαμε να προσθεθεί μια διάταξη έτσι ώστε οι οριακές τιμές της οδηγίας να επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να λάβουμε υπόψη και τις ε, επιστημονικές γνώσεις. Επίσης θα θέλαμε να ε, έχουμε ένα ε, σχέδιο ελαχιστοποίησης τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει ε, σχέδιο υποκατάστασης. Τέλος, θα ήθελα να σας μιλήσω για τις μακροχρόνιες προοπτικές για να μειώσουμε τον καρκίνο στην εργασία. Δεν υπάρχει μεθοδολογία στην ε, ίδια την οδηγία για το πώς να αντιμετωπίσουμε τις καρκινογόνες ουσίες. Θα πρέπει να αναπτυχθεί σε σχέση και με τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης γιατί βασιζόμαστε σε μία ανάλυση κόστους ωφελίας αποκλειστικά μέχρι τώρα. Είναι δηλαδή ε, σαν μία ρόδα που γυρίζει, σαν ένα μεγάλο στίχημα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό τη στιγμή που μιλάμε για οριακές τιμές και επαγγελματικά στοιχεία και για την ανθρώπινη υγεία βεβαίως πρωτίστως. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η τέταρτη εμπειρογνώμων, η Ρεμπέκα Σμιθ από το Business Europe. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Καταρχήν να υπογραμμίσω ότι συμφωνούμε για την πρόληψη των επαγγελματικών εκείνων, αυτό είναι και υπέρ των εργαζομένων της κοινωνίας αλλά και των επιχειρήσεων. Επίσης, αν είναι δεσμευτικά τα όρια έκθεση σε νοσιακό επίπεδο, θα υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και για την προστασία ως Business Europe λοιπόν. στηρίζουμε ως γενικό κανόνα τις περιορισμένες αναθεωρήσεις των παραρτημάτων 1 και 3 της οδηγίας για τα καρκινογόνα και μεταλλαξιογόνα και είμαστε υπέρ των δεσμευτικών ορίων έκθεσης. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για να θεσπιστούν πρόσθετες τιμές. Πρώτον, πιστεύουμε ότι η διαδικασία πρέπει να στηρίζεται σε ε, σωστές επιστημονικές πληροφορίες. Ε, ακούσαμε τι επιστημονικές πληροφορίες και δεδομένα υπάρχουν. Ε, πρέπει να είναι αξιόπιτα στα τα στοιχεία Πρέπει επίσης να στηριχθούμε σε μελέτες βιωσιμότητας, ε, σε τεχνικό επίπεδο, επιστημονικό επίπεδο και να δούμε και τις μελέτες αντικτύπου. Οι ουσίες που έχουν αποδειχθεί και ταξινομηθεί ως καρκινογόνες θα είναι αυτές που θα προσθεθούν στο παράρτημα της οδηγίας γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι οδηγία για, τα, για τους καρκινογόνους παράγοντες, οπότε έχει νόημα. Επίσης πιστεύουμε ότι δεν έχει νόημα να βάλουμε ένα το ε, αριθμητικό στόχο 50, 100, 200 πρόσθετα όρια δεσμευτικά μέχρι το 2020 χωρίς σαφή ιεράρχηση, θέση προτεραιοτήτων σχετικά με τους παράγοντες για τους οποίους χρειάζεται δεσμευτική τιμή. Ίσως είναι χρήσιμο να πούμε δύο λόγια για τη διαδικασία και να την εξηγήσουμε. Ξέρουμε όλοι ότι η Κομισιόν είναι εκείνη που κάνει την πρόταση για τις τιμές όρια, αλλά μετά γίνονται πολλές δουλειές, διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους, όλα αυτά γίνονται πριν. Και είναι σημαντικό να το θυμηθούμε αυτό εδώ. Θα γνωρίζετε ίσως ότι οι εργασίες αρχίζουν τουλάχιστον σε ενωσιακό επίπεδο στην Επιστημονική Επιτροπή για τα όρια επαγγελματική έκθεσης, ΣΚΟΕΛ, που σκοπό έχει να δει τα επιστημονικά δεδομένα αν η τιμή όριο είναι στα πλαίσια των υφισταμένων τεχνικών μέτρησης και μας δίνει και feedback από πολλούς εμπλεκομένους ε, κυβερνήσεις, εργαζομένους, εκπροσώπους της βιομηχανίας. Μετά γίνεται η συζήτηση στην Γνωμοδοτική Επιτροπή και αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα στη διαδικασία γιατί αυτή η Επιτροπή, η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τρεις εκπροσώπους ε, κυβερνήσεων εργοδοτών εργαζομένων και ο ρόλος της είναι να δει αν οι προτινόμενες τιμές από τη ΣΚΟΕΛ, την Επιστημονική Επιτροπή, πληρούν τα κριτήρια κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο, δηλαδή και βιωσιμότητα, εφικτότητα. Και οι προηγούμενοι ομιλητέ μίλησαν για ανάλυση κόστους οφέλους, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Βέβαια δεν θα βάλουμε σε ίδια μοίρα το κόστος για τη βιομηχανία και το κόστος στην ανθρώπινη υγεία. Πιστεύουμε όμως πολύ στη βιωσιμότητα, στο κατά πόσο είναι εφικτά όλα αυτά. Να φροντίσουμε ότι η βιομηχανία μπορεί να εφαρμόσει τις, ε, τα όρια έκθεσης και να προστατεύσει τους εργαζομένους. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Τώρα, η Συμβουλευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή καμιά φορά υπάρχει ξεκάθαρη συμφωνία μεταξύ των τριών μερών, καμιά φορά δεν συμφωνούν. Ε, αλλά το έργο της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα όρια τιμών που προτείνει τουλάχιστον στις γνωμοδοτήσεις της ήδη είναι μια καλή στέρεα βάση και δίνουν μια γενική προσέγγιση για να ακολουθήσει η Κομισιόν. Και χαιρόμαστε που στην πρόταση της Κομισιόν φαίνεται ότι ακολουθούν την, ακολουθεί την ε, γνωμοδοτική, τη συμβουλευτική αυτή επιτροπή. Είναι αλήθεια ότι όλες αυτές οι διαδικασίες μπορεί να είναι κάπως χρονοβόρες, συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή, γιατί παίρνει χρόνο μέχρι να ενημερωθούν οι τιμές για τα όρια και καλό είναι να βρούμε απλούσταρες, ε, ταχύτερες διαδικασίες για να αναπροσαρμόζουμε σε νοσιακό επίπεδο τα όρια επαγγελματικής έκθεσης, τις σχετικές τιμές. Όμως δεν πρέπει να γνωρίσουμε και να, δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουμε από τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί, γιατί χρειάζονται, να, ώστε να υπάρχει μια γενικότερη προσέγγιση που θα οδηγήσει σε συνένεση των εμπλεκομένων. Πρέπει να πούμε επίσης ότι είναι γνωστό ότι θα υπάρχει δεύτερο και τρίτο κύμα προτάσεων και αυτά που είπα αφορούν και αυτές τις προτάσεις. Οι προϋποθέσεις που έθεσα δηλαδή για να θεσπιστούν ε, δεσμευτικά όρια ισχύουν για όλα τα κύματα Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες σε επιμέρους κλάδους της ε, βιομηχανίας σχετικά με ορισμένες τιμές όριο που έχουν προταθεί ή τη συμπερίληψη κάποιων παραγόντων στην οδηγία για τα καρκινογόνα. Γνωρίζετε βέβαια ότι υπήρξε μακρά συζήτηση σχετικά με την μικρή κρυσταλλική πυρητία και αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί και βλέπουμε ότι η επιστημονική κοινότητα αναλύει με διαφορετικό τρόπο την ουσία αυτή. Δηλαδή, ακόμα σε ένα βαθμό υπάρχει έλλειψη συνένεσης πάνω σε αυτή την ουσία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες σε κάποιους τομείς ε, σχετικά με το αν πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία για τα καρκινογόνα και πρέπει να Αναφέρουμε επίση ότι δεν πρόκειται μόνο για τις οριακές τιμέ, αλλά και για την εφαρμογή και των άλλων μέτρων που προβλέπει η οδηγία. Ε, μιλάω εδώ για την ιεράρχηση των μέτρων, δηλαδή να δούμε αν χρειάζονται μέτρα υποκατάστασης, αν στο χώρο εργασίας θα πρέπει να υπάρχει κλειστής διαδικασίας προσέγγιση σε κλειστό σύστημα. Επίσης γνωρίζομαι και εσείς γνωρίζετε νομίζω και συμφωνούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν αναφέρεται στο, στη συμφωνία ε, πολλών κλάδων ε, και υπάρχει εδώ ε, αναφορά στην ε, πυρητεία. νομίζομαι ότι είναι καλό που αναφέρεται. Αναφέρεται και στη συνεργολογική σκέψη ότι η συμφωνία είναι συμπληρωματική. Και θα πρέπει να δούμε αυτή η συμπληρωματικότητα πώς θα λειτουργήσει στην πράξη η συμφωνία σε σχέση με την οδηγία. Δηλαδή θα μπορεί η συμφωνία να έχει ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια της για να εφαρμόζει και τις ε, οριακές τιμές ε, και τις ε, διατάξεις για την επικινδυνότητα. Έχουμε κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τις οριακές τιμές που θεσπίστηκαν για τις σκόνες σκληρού μετάλλου. Υπάρχουν θέματα δηλαδή για, τα, για το κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστούν. Έχουμε πληροφορίες από κάποιους τομείς ότι κάποια μηχανήματα, χειροκίνητα που χρησιμοποιούνται σε κάποιους τομείς, όπου υπάρχει σκόνη σκληρών ξύλων, ότι είναι δύσκολο να κατέβουν κάτω από την σημερινή οριακή τιμή. Παρά τα τεχνικά οργανωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Ε, είναι θέμα μηχανήματος. Αυτό εννοώ όταν λέω τεχνική εφικτότητα. Ε, ε, τα τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή των οριακών τιμών και των γενικότερων μέτρων. Έχει γίνει συζήτηση για το χρώμιο 6, το εξασθενές χρώμιο. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ζήτημα στη συζήτηση του Συμβουλίου τώρα και όπως είπε και η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία μπορεί να υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ε, ένα χρονικό διάστημα για να αναθεωρηθεί η τωρινή οριακή τιμή ε, παράλληλα είναι σημαντικό να δούμε τους διάφορους τομείς ε, τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας που χρησιμοποιούν το εξασθενές χρώμιο και τι σημαίνει αυτό στον ανασχεδιασμό των παραγωγικών διαδικασιών, κλειστά συστήματα κλπ. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι αν και μπορεί να χρειαστεί να καθοριστεί ένα χρονικό όριο για την αναθεώρηση, θα πρέπει να είναι πολύ ισορροπημένη η προσέγγιση μας εδώ εν συμπεράσματι, αν και έχουμε κάποιες ε, επιφυλάξεις ό,τι αφορά κάποιες οριακές τιμές που προτείνονται ή με τη συμπερίληψη κάποιων παραγόντων στην οδηγία, ε, σας ενθαρρύνουμε να προσπαθήσετε να μείνετε όσο πιο κοντά γίνεται στην πρόταση της Κομισιόν. Και γιατί το λέω αυτό. Όπως είπα και πριν, η Γνωμοδοτική Επιτροπή συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό και εκεί εκπροσωπούνται εργοδότες εργαζόμενη κυβέρνηση. Στηρίζονται σε ε, επιστημονικές αποδείξεις, στοιχεία και υπάρχει ευρεία στήριξη και μεταξύ των κρατών μελών από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να ανοίξουν τα άρθρα της οδηγίας. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η αναθεώρηση να περάσει γρήγορα, να θεσπιστούν οι οριακές τιμές δεσμευτικές στην οδηγία και νομίζουμε ότι αν αρχίσουμε πιο περίπλοκη συζήτηση για αλλαγή των άρθρων, αυτό θα επιβραδύνει τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην πρόταση της Κομισιόν αυτή καθ' αυτή για να πάμε γρήγορα και να, να έχουμε γρήγορη πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εμπειρογνώμονές μας. Πριν δώσω το λόγο στη Μαρίτα τώρα, επιτρέψτε μου μια απόλυτα προσωπική παρατήρηση. Με εκπλήσει πόσο εύκολα συζητάτε για τη σχέση μεταξύ κόστους και ωφέλειας. Έχω καρκίνο και αν είναι κανείς ε, θύμα μιας τέτοιας εκτίμησης κόστους ωφέλους αισθάνομαι κάπως άβολα αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις αλλά θα επανέλθω σε αυτές θέλω να δώσω τον λόγο στη Μαρίτα θα μιλήσω σουηδικά Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για όλα αυτά για τα οποία μας ενημερώσατε. Είναι σαφές από αυτά που μόλις είπε ο πρόεδρός μας ε, Τόμας Έντολ, είναι ότι όλοι έχουμε μια πολύ προσωπική σχέση με τον καρκίνο και Αυτό ισχύει για όλες τις ιδιαίτερα διαδεδομένες ασθένειες. Ε, ε, είναι κάτι που μας θίγει ως άτομα. Δεν είμαστε μόνο πολιτικοί, ε, είμαστε και ανθρώπινα όντα και αυτό είναι σαφές στην εργασία που κάνουμε τώρα. Και επηρεάζει και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καρκινογενείς. Τώρα κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρατε. που είναι πολύ σημαντικά για μας. Είναι οι άξονες της δράσης μας. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι έχουμε 102.500 θανάτους στην Ευρώπη το χρόνο είναι τρομερός αριθμός αυτός. Είμαστε το ε, υγιέστερο, πλουσιότερο τμήμα του κόσμου. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της ε, προσπάθειας αντιμετώπισης των σοβαρών ασθενειών. Αυτός ο αριθμός, 102.500 άτομα, θα είναι ακριβώς και η βάση για τις προτάσεις μας, η μείωσή του. 53% όλων των επαγγελματικών θανάτων, των θανάτων δηλαδή που σχετίζονται με την ε, επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλονται στον καρκίνο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που επίσης ε, θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οικονομικά και άλλα συμφέροντα που παίζουν ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Άρα πάντα χρειάζεται να έχουμε φιλόδοξους στόχους να δίνουμε φιλόδοξους στόχους και για τα κράτη-μέλη. Δεν έχει έννοια να αποφασίσουμε κάτι το οποίο να μην είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα μισά, ας πούμε, κράτη-μέλη. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι έχουμε ιδιαίτερα υψηλέ προσδοκίες ως Επιτροπή. Διότι όλοι γνωρίζουμε, βεβαίω, ότι οι προτάσεις μας πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Και αυτό το γνωρίζουμε. Και πρέπει να είναι σταδιακή η προσέγγιση Βέβαια δεν θα θέλαμε. Θα θέλαμε να υπάρξει ραγδαία πρόοδος για την αντιμετώπιση αυτών των καρκινογενών, αλλά πρέπει να έχουμε ευρία υποστήριξη, άρα η φιλοδοξία μας πρέπει να συνδυάζεται με αποτελεσματικότητα. Όλα όσα μας παρουσίασαν για τα, τις καρκινογόνες ε, στον τόπο εργασίας οι ερευνητές είναι πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά. Παράλληλα όμως πιστεύω ότι η εργασία μας θα επηρεαστεί και από ορισμένα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων γιατί υπάρχουν ε, οικονομικές ε, επιπτώσεις, υπάρχουν ε, διχογνωμίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Υπάρχουν διαφορές και μεταξύ κρατών μελών. Σε ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζονται οι καρκινογόνες στον τόπο εργασία και στην κοινωνία γενικότερα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Σε άλλα κράτη-μέλη από την άλλη μεριά έχει σημειωθεί μικρότερη πρόοδος. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, ότι είναι άνηση λοιπόν η αποτελεσματικότητα της μεταχείρισης. Εμείς ως Επιτροπή λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει μέσω της δράσης μας να βοηθήσουμε τους βραδιπορούντες να καλύψουν αυτή την καθυστέρηση. Τούτων λεχθέντων να τονίσω ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους με πολύ προσωπικό τρόπο. Είναι ένα θέμα γενικού συμφέροντος, αλλά είναι ένα θέμα και προσωπικού συμφέροντος όλων μας και καθενός εξημών. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας. Έμαθα ορισμένα νέα πράγματα από τις παρουσιάσεις σας. Βεβαίω ε, είχα και ε, γνώσεις αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα από κοινού, ούτως ώστε, να έχουμε ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα. Να τονίσω κάτι το οποίο έχει αναφερθεί από διάφορους ομιλητές. Ε, το είπατε στις ομιλίες σας ότι υπάρχει και διάσταση φίλους στα θέματα αυτά. Γιατί μέχρι στιγμής ορισμένες μελέτες για τον καρκίνο το αγνοούν το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνεται τώρα η διάσταση του φύλου. Είναι σημαντική και αυτή και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μαρίτα. Οι σκιώδεις συζητητές. Κλοντ Γολέμο πρώτος. Κλοντ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ θα έπρεπε να πω ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με υψηλή, υψηλότατη τεχνολογία, τεχνολογία εχμής, δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Μιλήσαμε για τη σχέση μεταξύ υγείας και κόστους συμμόρφωσης. Υπάρχουν και δεοντολογικά ζητήματα. Θα ήθελα όμως να μου πείτε Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό τον υπολογισμό. Είναι τα ίδια στοιχεία που έχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείε ή όχι. Επίσης έχει σημασία η εκδήλωση καρκίνου μετά την έκθεση στην εργασία, μετά την περίοδο εργασίας. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε τους εργαζόμενους. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για το βιομηχανικό τομέα, αλλά και στις υπηρεσίες. Όχι με καθαρά προϊόντα ή σωματίδια. Θυμάμαι ότι είχα ασχοληθεί με τις υπηρεσίες καθαρισμού και είδα ότι έρχονταν σε επαφή με ένα μείγμα διαφορετικών προϊόντων και ενώσεων και δεν ήξεραν τι ε, προκαλούν. Η κυρία Σνάιντερ μίλησε και για τον τομέα των κομμωτηρίων. Εδώ φτάσαμε σε συμφωνίες και ελπίζω η Επιτροπή να συμμορφωθεί με αυτές τις συμφωνίες, να είναι λίγο πιο συνεπής από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι οριακές τιμές στα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο ανταγωνισμού, αλλά γιατί ό,τι λειτουργεί σε μια χώρα να μην λειτουργεί και σε μια άλλη. θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση εκ του να μας απασχολεί η υγεία των εργαζομένων πρωτίστως, αλλά και να είμαστε και ρεαλιστές ως προς το εφικτό. Δεν έχει νόημα να ορίζουμε στόχους από τις οποίους θα υπεκφύγουν πολλοί. Μιλάμε για 100.000 ενώ στον τομέα των ατυχημάτων στις οδικές αρτηρίες οι θάνατοι ανάρχονται στις 25.000. Θα πρέπει και εκεί να γίνει ε, πρόληψη, αλλά και εδώ θα πρέπει να κάνουμε το αντίστοιχο. Να έχουμε τα νομικά μέσα, μέσω οριακών τιμών, αλλά θα πρέπει να γίνει και πρόληψη και επαγρύπνηση όπως γίνεται σε επίπεδο ε, νέψη. Πρόκειται για έναν τομέα που ορίζει πρακτικές που ορίζονται από τους εργαζόμενους επιτόπου. Αυτά τα μέσα θα μας βοηθήσουν για να μας καθοδηγήσουν, για να μειωθεί η εκδήλωση επαγγελματικού καρκίνου ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Ίσως αυτά που κάνουμε, ίσως να μην βλέπετε τις ε, διαφάνειες, ε, αλλά βοηθάνε παρόλα αυτά. Δεν είναι εδώ η Ανθέα Μάκιντάρ, είναι κανείς άλλος. Εσείς. Ποιος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αντικαθιστώ την εισηγήτριά μας, την κυρία Μάκιντάρ. Σας ευχαριστώ όλους. Για να καταλήξουμε σε συμφωνία πρέπει να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Γενικά συμφωνώ ότι πρέπει να προσταθούν και άλλες ουσίες στον κατάλογο καρκινογόνων του 2004. Πρέπει να είναι προτεραιότητα η αποφυγή επαγγελματικών καρκίνων. Είναι προς το συμφέρον όλων και εργοδοτών και εργαζομένων. Και θεωρώ ότι τα δεσμευτικά όρια σε ενωσιακό επίπεδο μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε ο κλάδος να εργάζεται σε συνθήκε ε, θεμητού ανταγωνισμού και φυσικά να υπάρξει και προστασία των εργαζομένων παντού στην Ένωση. Η διαδικασία αυτή Πρέπει να βασιστεί βέβαια στην επιστημονική γνώση, αλλά πρέπει να υπάρχει και τεχνική ε, εφαρμοσιμότητα και να έχουμε υπόψη και την κοινωνικονομική πλευρά του θέματος. Να, είμαστε, να βασιζόμεθα στα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και να μην ορίσουμε αυθαίρετα ανώτατες τιμές, γιατί αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να θίξουμε την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και άρα και την απασχόληση θα μπορούσα να συμφωνήσω με την αναθεώρηση των ε, παραρτημάτων, αλλά όχι το κείμενο της ομιλίας και προσβλέπω στη συνεργασία με τους σκιώδεις ε, τους επόμενους μήνες και την εισηγήτρια. Δεν. είναι. Πάτρικ όχι. Καρίμα Ντελή, για τους πράσινους, όχι. Ούτε ζητεί άλλο το λόγο. Η FTD το ίδιο. Σουέλ Μελέν. Τι είναι; Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους προγνώμενους που ήρθαν ε, να συμβάλλουν στην ενημέρωσή μας. Χαίρομαι που άκουσα τους εκπροσώπους της οργάνωσης ε, ΤΟΥΙ. Ευχαριστώ λοιπόν που άκουσα για τη δική σας γνώμη. Λοιπόν, μερικές προτάσεις για, ε, το πού θα καταλήξουμε. Είναι πραγματικά σκανδαλώδες να μιλάμε για κόστος όφελος. Καλύτερα λοιπόν στο κείμενο να μιλήσουμε μόνο για το κόστος γιατί είναι το κόστος των επιχειρήσεων. Και το κόστος για τις επιχειρήσεις ε, πολύ συχνά μειώνει την πρόληψη. Και η πρόληψη πρέπει να είναι ο στόχος μας. Να προλαμβάνουμε και να προβλέπουμε. Γιατί ξέρετε ότι η περίοδος έκθεσης ε, παίζει μεγάλο ρόλο και επίσης υπάρχει και η, η περίοδος επόασης των ασθενειών. Το κόστος οφείλεται στις ε, ιδιαίτερα περίπλοκες και δαπανηρές ε, επενδύσεις. Ε, όταν, για παράδειγμα, αναφερόμεθα στις μηχανές για την καταργασία του ξύλου που χειρίζονται οι ίδιοι εργαζόμενοι, καταλαβαίνετε και ξέρετε ότι και οι εργαζόμενοι ήδη αλλά πολλές φορές και οι γυναίκες τους που καθαρίζουν τις στολές τους. Είναι κόστος, που αφορά και την οικογένεια και το κόστος επίσης ε, της απώλειας εργατοημερών και το κόστος για την κοινωνική ασφάλιση. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες πλευρές του κόστου. Του κόστους. Αλλά το κόστος συνολικά είναι ουσιώδες. Δεν είναι σωστό όμως να μιλάμε για σχέση κόστους ωφελίας. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το κόστος βράχη, μέσο και μάκρο πρόθεσμα. Τώρα βέβαια η εκπρόσωπος της οργάνωσης Business Europe είπε να διατηρήσουμε το κείμενο γιατί έτσι θα εγκριθεί ευκολότερα. Α, θα μπορούσα να το κατανοήσω αλλά ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στο κείμενο αυτό κάποια στοιχεία πρόληψη, δηλαδή να αναφερθούμε στις ουσίες αλλά όχι σε όρια. Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Αυτή είναι η πρόταση που έχω να κάνω και σας ευχαριστώ πολύ. Χουκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ε, ειδικού για την ενημέρωση που μας έκαναν και ίσως μπορούμε να μαλώσουμε για την οδηγία, για την απόσπαση ή για άλλες οδηγίες γιατί και η διαφωνία είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Όταν όμως μιλάμε για καρκινογόνα και ε, μεταλλαξιογόνα στον τόπο εργασίας πρέπει να μιλάμε με μία φωνή. Διότι αν ένας εργαζόμενος ακούσει ότι έχει ε, καρκίνο και μάλιστα επαγγελματικό τότε δεν μετράει τίποτα άλλο, ούτε τα κέρδη της επιχείρησης, ούτε η αύξηση της αποδοτικότητας, ούτε οι καινοτομίες, ούτε η αποζημίωση. Το μόνο που μετράει είναι η υγεία και η ζωή του εργαζομένου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, η ύψιστη άξια. Και επειδή είμαι γιατρός, με σχεδόν 40 χρόνια επαγγελματική πείρα, έχω δει ε, δεκάδες τέτοιες διαγνώσεις και ξέρω τι τραγωδία είναι. Και από ιατρικής πλευράς μπορώ να πω ότι μια διάγνωση καρκίνου δεν είναι καταδίκη σε ναι. θάνατο, γιατί ένα μεγάλο ε, ε, ποσοστό των καρκίνων είναι ιατή με την προϋπόθεση ότι θα αναγνωριστούν και θα διαγνωστούν έγκαιρα. Όμως, μια σημαντική πληροφορία είναι ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του καρκίνου και το καλύτερο φάρμακο για τον καρκίνο είναι η προφύλαξη. Και φοβούμε ότι αν και οι διατάξεις στα κράτη-μέλη είναι διαφορετικές, παρόλα αυτά δεν τηρούνται και δεν εφαρμόζονται. Εδώ μιλάμε για πάνω από 100.000 κρούσματα θανάτων κατέτος. Άρα 100.000 ε, ε, άνθρωποι εξαφανίζονται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη κάθε χρόνο. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Ε, μου άρεσε η θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων που δεν μίλησε καν για κόστος και όφελος. Είπε ότι το μόνο που μετράει είναι η ζωή και η υγεία των εργαζομένων. Γιατί αν δεν τα αυτά θα είμαστε μια Ευρώπη αρνητικών αξιών. Υπάρχουν επίσης και τρομακτικές πληροφορίες. Ακούμε ότι ε, το προσωπικό καθαρισμού, οι κομμωτές και κομμότριες είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις ουσίες. Φανταστείτε τι γίνεται σε μια βιομηχανία. Σε κάποιες χώρες, κυρίως στην κεντρική και ανατολική κυρίως Ευρώπη, αυτά τα πρότυπα, οι τιμές δεν τηρούνται καθόλου ούτε υπάρχει κάποιο κεντρικό μητρό ή αρχείο όπου θα καταγράφονται οι κίνδυνοι αυτοί. Γι' αυτό το λέω και το, και το τονίζω. Ε, εδώ πρέπει να δράσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα και οι ευρωπαϊκές οριακές τιμές θα πρέπει να θεσπιστούν το ταχύτερο δυνατόν και να τηρούνται και στην πράξη. Μπορεί, όπως είπα, να διαφωνήσουμε σχετικά με το πόσο, κατά πόσον θα προσαρμόζονται στα δεδομένα της κάθε χώρας. Όμως θα πρέπει να θεσπιστούν και να ισχύσουν, διότι εδώ παλεύουμε για τις θεμελιώδεις μας αξίες και για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων, που όπως είπαμε είναι η ανώτατη ύψιστη αξία, πέρα από κόστος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Καρίμα Ντελή δεν μπόρεσε να παρευρεθεί δυστυχώς. Ε, θα προσπαθήσω εγώ να παρουσιάσω κάποια σημαντικά θέματα για την ομάδα μας. Είμαστε ευτυχείς διότι επιτέλους βλέπουμε να κινείται η συζήτηση και η διαδικασία. Είχαμε προτάσεις για πολύ καιρό σε αυτό το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία και αυτό, είναι, ε, αυτό αφορά ιδιαίτερα τα καρκινογόνα που επηρεάζουν τόσα εκατομμύρια ανθρώπων. Ε, στηρίζουμε λοιπόν πολύ την εξέλιξη σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, θέλουμε κάποιες αλλαγές και βελτιώσεις. Θέλουμε συγκεκριμένα να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής για να συμπεριλάβει και άλλες επικίνδυνες ουσίες για την αναπαραγωγή. Το είπαν κάποιοι συνάδελφοι και θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες για να δούμε τι μπορεί να, ακόμα να γίνει. Εδώ. Επίσης θέλουμε να μειωθούν τα μέγιστα, οι μέγιστες ποσότητες, γιατί όπως αναφέρθηκε, αν ε, ε, ε, ότι σε κάποια κράτη-μέλη είναι δυνατόν να ισχύουν αυστηρότερα πρότυπα. Καλό είναι λοιπόν οι βέλτιστε αυτέ πρακτικέ να επεκταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε την καλύτερη προστασία όλων των εργαζομένων τη Ένωση. Τέλο, ο τομέα των υπηρεσιών πρέπει και αυτό να συμπεριληφθεί, γιατί ε, είναι πολλέ οι γυναίκε που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και οι οποίες αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία τους. Και αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σημείο για μας. Εξ ονόματος της συναδέλφου Καρή Μαντελή πρέπει να πω ότι προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική και παραγωγική συζήτηση. Ο κύριος Λάμπρος Φουντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για τη συζήτηση αυτή και θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Συμφωνώ με τη μείωση των τιμών στις καρκινογόνες ουσίες και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτές τις ουσίες που έχει αποδειχτεί ότι κάνουν μεγαλύτερο κακό. Παράλληλα όμως θα ήθελα να προτείνω ότι πρέπει να γίνει και μια καμπάνια για μέτρα προστασίας των εργαζομένων και η εφαρμογή τους από τους ίδιους εργαζόμενους, οι οποίοι είτε από άγνοια, είτε από διαφορία ή και λένε ότι, λέγοντας ότι δεν θα συμβεί αυτό σε μένα, έρχονται αντιμέτωποι με την ασθένεια. Ο καρκίνος που συνδέεται με την εργασία είναι ένα ύπουλος καρκίνος, διότι αρχίζει να εκδηλώνεται πολλές φορές μετά το πέρας του εργασιακού βίου. Ε, Επίση, είναι λάθο να μιλάμε για κόστο και όφελο όταν μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτήμητη. Ευχαριστώ. So, dann stehe ich selber auf der Redeliste. Πότε τώρα να μιλήσω και εγώ ίδιος. Να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Και το κάνω συνειδητά πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θεωρώ ότι τρία θέματα πρέπει να αναφερθούν ακόμη σε σχέση με τον καρκίνο. Πρώτον, με εκνευρίζει κάπως το ότι δεν έχουμε ακόμη επαρκή στατιστικά στοιχεία. Ξέρω από ίδια εμπειρία ότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία είναι σε φάση εκπόνησης ένα εθνικό μητρό καρκίνων. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε τα αίτια. Ιδιαίτερα οι ιατροί, οι ογκολόγοι λένε ότι δεν ξέρουν ακριβώς το αίτιο του 80% των καρκίνων. Δεν έχει αποδειχθεί σαφώς από ιατρική άποψη η προέλευση των καρκίνων. Δεύτερον, με ανησυχεί το ότι όλο και συχνότερα νέοι άνθρωποι ε, ε, παθαίνουν καρκίνο. Ξέρω ότι πολλές φορές η χρήση προστατευτικών μέσων, για παράδειγμα ακουστικά, μάσκες και άλλος τέτοιος προστατευτικός εξοπλισμός δεν θεωρείται έτσι μοντέρνος από τους νέους και δεν τα βάζουν. Δεν είναι δυνατόν όμως να γίνονται αυτά τα πράγματα. Μήπως θα έπρεπε από τη μία να κάνουμε μια ενημερωτική εκστρατεία και από την άλλη να επιμένουμε στην αυστηρότερη εφαρμογή των κανονισμών για τον προστατευτικό εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε για λόγου έτσι ότι δεν γουστάρουν να μην φοράνε τον προστατευτικό εξοπλισμό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να το σκεφτούμε. Και το τρίτο. Από προσωπική και πάλι εμπειρία γνωρίζω ότι όπως ανέφερε και προηγούμενο ένας συνάδελφος Ξέρω λοιπόν ότι σήμερα γνωρίζουμε ότι ε, πρέπει να κάνει κανείς πάρα πολλές ε, εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν έχει τον ε, αν έχει καρκίνο και επίσης η μέθοδοι για την διάγνωση του καρκίνου και για ε, την εκτίμηση αν έχει υπάρξει θεραπεία μετά από πέντε χρόνια είναι πολύ ανομοιογενείς αυτές οι ε, μέθοδοι και τα κριτήρια. Αυτές είναι οι τρεις ερωτήσεις και κάνω αυτές τις ερωτήσεις για να μας ε, πούν τη γνώμη τους οι δήμονες και η δική μας εμπειρογνώμονη Μαρίτα και η Κομισιόν. Οπότε πρώτα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν η Τερέζα Μουτίνιο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την ε, παρουσίαση των ε, εμπειρογνωμόνων σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Η πρόταση της Επιτροπής του παρελθόντος Μαΐου είναι φιλόδοξη γιατί θεωρούμε ότι έχει επιτελεστεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη βελτίωση και τη προστασία των εργαζομένων ως προς την υγεία και ασφάλειά τους στο χώρο εργασίας. Ευπρόσδεκτη λοιπόν αυτή η πρόταση και μετά από μία ε, ευρεία διαβούλευση και με επιστημονικούς φορείς έγινε δεκτή αυτή η έκθεση. Και μετά την ε, τριμερή συμβουλευτική επιτροπή, την γνωμάτευση της τριμερούς συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας. Επίσης ε, έγινε και μία εξωτερική ανάθεση ε, διενέργειας μιας μελέτης για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας. Και φτάσαμε και στις ε, οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που βλέπετε στην τελική μας πρόταση. Θεωρώ ότι οι δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης ε, είναι απαραίτητες και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους και κυρίως για τους εργοδότες, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων. Αλλά και οι άλλες αρχές της οδηγίας ισχύουν δηλαδή μείωση της έκθεσης κατά το ελάχιστο δυνατόν. Θα δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου εάν θέλετε λεπτομεριακή σχολιασμό ορισμένων ζητημάτων και μετά θα επανέλθω στα ερωτήματα του Προέδρου. Ευχαριστώ Τερέζα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Ένα από τα βασικά ζητήματα που με απασχολεί είναι ε, ο σχεδιασμός της οδηγίας για τις καρκινογόνες ουσίες. Μιλάμε για οριακές τιμές καταρχήν, αλλά η οδηγία έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο από τις ουσίες που καταγράφονται. Ε, και αντικατοπτρίζει τη σημασία του ζητήματος. Φτάνουμε λοιπόν σε οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης στα παραρτήματα, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να απαλείψουμε την έκθεση εκεί που γίνεται. Διαφορετικά θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την έκθεση ή να μην υπάρχει καθόλου έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, πέρα από αυτές που αναγράφονται στα παραρτήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί, γιατί οι περισσότερες καρκινογόνες ουσίες δεν μπορούν να έχουν κατώτερη οριακή τιμή. Δεν μπορεί να οριστεί κατώτερη τιμή γιατί ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδηγία έχει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Εδώ μιλάμε για χημικές ουσίες που δεν μπορούν να αποτιμηθούν ως προς ένα κατώτατο όριο. Γιατί, όπως γνωρίζετε, ε, πολλές ουσίες έχουν οριακές τιμές αλλά εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα σε θέματα ε, αναπαραγωγικής τοξικότητας. Ως προς τις ενδεικτικές οριακές ε, τιμές που εμπίπτουν σε μία άλλη οδηγία, θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο δεσμευτικά αυτά τα μέτρα. Εμείς δεν συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη θεωρώ ότι θα πρέπει και οι ενδεικτικές οριακές τιμές να μεταφερθούν από τα κράτη-μέλη. Και εδώ μιλώ για την οδηγία χημικών ουσιών. Άρα δεν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο και οι ενδεικτικές ε, οριακές τιμές. Ως προς το εξασθενές χρώμιο θα ήθελα να πω ότι από τις 13 ε, ουσίες αυτής της ε, πρότασης το χρώμιο 6 είναι το μόνο σύμφωνα με το οποίο ε, το κόστος που ζητάμε που ενέχεται στις οριακές τιμές είναι πολύ χαμηλότερο από τα ευεργετήματα, γιατί ξέρουμε το χρώμιο 6 είναι μία ενεργός καρκινογόνος ουσία και στοιχεί στην Ευρώπη περισσότερο από ό,τι την ωφελεί. Γι' αυτό θέλουμε και να προβάλλουμε μία συνολική πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δώσατε και το λόγο. Εάν μου επιτρέπετε, θα επανέλθω στις δικές σας συγκεκριμένες ερωτήσεις. Χρειάζομαστε βελτιωμένα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν κάνει εξωτερική ανάθεση για μία μελέτη για να δούμε την βιωσιμότητα και το εφικτό το δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων για την έκθεση σε χημικές ουσίες. Πρόκειται για την μελέτη Haschem, η οποία τώρα βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ε, ληφθούν και μέτρα εποπτείας και επαγρύπνησης και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επικείμενη εκστρατεία υγείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού σε σχέση με τις επικίνδυνες ουσίες, την έκθεση για, ε, στις επικίνδυνες ουσίες. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ασχοληθούμε με επιμέρους θέματα έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τους νέους και ε, ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων που εκτίθενται σε καρκινογόνες ουσίες. Τώρα, ως προς τη διαθεσιμότητα στοιχείων, το πρώτο σας ερώτημα, Μίλησα για τον οργανισμό του Bilbao, ο οποίος θα ασχοληθεί με μία μελέτη για την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα κριτήρια διάγνωσης στα κράτη-μέλη και θα θέλαμε να σας επισύρουμε την προσοχή σε μια πολύ σημαντική έκθεση των υπηρεσιών της Κομισιόν εδώ και μερικά χρόνια, δηλαδή ένα δελτίο για διαγνωστικά κριτήρια, τα οποία θα μας βοηθούσαν να υπάρχει μια ευρύτερη πληροφόρηση σε σχέση με τις επαγγελματικές ασθένειες. Και τώρα οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταβάλουν προσπάθειες για να ενεργοποιήσουν ε, ένα μηχανισμό στατιστικών στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες το σχέδιο ΕΑΤΣ και μαζί με τη Eurostat θα αρχίσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για έναν απλοποιημένο κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών που θα την χάνουν των ίδιων κριτηρίων διάγνωσης στα κράτη-μέλη. Και για να βελτιώσουμε την κατάσταση βεβαίως όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος πάλι στους και στις εμπειρογνώμονες με τη σειρά. Όμως πρέπει να ακολουθήσουμε έναν κανόνα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προβλέψει σε αυτές τις περιπτώσεις ένα λεπτό χρόνο ομιλίας. Ε, βέβαια θα είμαι ανεκτικός η Λέσλι Ράστον. Ευχαριστώ. Με ενδιαφέρον άκουσα τις πολλές και διάφορες γνώμες. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης να ακούσουμε και την, τη σκοπιά των ασθενών και συμφωνώ ότι το έγγραφο της Κομισιόν δεν πιάνει και αυτή την πτυχή και τον αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά σε όλη την οικογένεια. Είναι δύσκολο να κοστολογηθούν τέτοια πράγματα. Όποια αδρά στοιχεία Υπάρχουν κάποια αδρά στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε, αλλά το κόστος το κοινωνικό είναι τεράστιο. σίγουρα επειδή θα, αυξηθούν και οι καρκίνοι και οι επαγγελματικοί παρόλο που πολλοί επιβιώνουν. Εγώ χαιρετίζω τις προσπάθειες που άρχισαν και θα συνεχιστούν και στη βιομηχανία και μεταξύ των εργαζομένων ώστε να μείνει ο κόσμος στην εργασία. Κάτι που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε τους ανθρώπους που είχαν πάθει καρκίνο και να φροντίσουμε να δουλέψουν μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Και βέβαια τα όρια συνταξιοδότησης στην Ευρώπη ε, γίνονται όλο και ψηλότερα. Σας ευχαριστώ. Η Έλκε Σνάιντερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω ε, στις δραστηριότητες ε, της ΩΣΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρκινογόνων εμείς ε, κάνουμε μια μελέτη, όπως είπε και η Λέσλη για την επιστροφή στη δουλειά καρκινοπαθών. Έχουμε για παράδειγμα μελέτες ε, περιστατικών στις επιχειρήσεις για να δούμε ποια ε, θέματα προέκυψαν σε επίπεδο επιχείρησης. Παίρνουμε συνεντεύξεις από ανθρώπους που τρέχουν τέτοια προγράμματα για να γυρίσουν οι καρκινοπαθείς στη δουλειά τους και ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εμπόδια στην επιτυχή επιστροφή. Ε, για τις δραστηριότητες της εκστρατείας, ε, μια προτεραιότητα είναι η πρόληψη και μια ομάδα προτεραιότητας είναι οι νέοι εργαζόμενοι. Θα τα ε, δούμε λοιπόν τα θέματα αυτά στις μελλοντικές δραστηριότητες. για την έρευνα ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη εφικτότητας για να τρέξει πια η πιλωτική φάση σε όλη την Ευρώπη ή σε κάποια κράτη-μέλη. Και ίσως να αποκομίσουμε καλύτερη εικόνα για τον αριθμό των ε, εργαζομένων και οι ομάδες οι ευάλωτες είναι σημαντικές και οι γυναίκες. Έγιναν κάποιες μελέτες σχετικά με την έκθεση των γυναικών εργαζομένων κυρίως στους καρκινογόνους παράγοντες. Ε, κάποιοι παράγοντες συζητούνται. Γιατί ορισμένοι καρκινογόνοι παράγοντες είναι πολύ σημαντική για τις γυναίκες γιατί η έκθεση αυξάνεται. Ευχαριστώ. Ε, ο Τόνι Μόσου. Ευχαριστώ. Να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Γιατί θέλουμε στόχους για αυτές τις 50 καρκινογόνες μέχρι το 2020. Αυτή είναι η δέσμευση της Επιτρόπου Τάισεν. Γιατί οι 50 χειρότερες καρκινογενείς θα καλύψουν το 80% των περιπτώσεων έκθεσης στον τόπο εργασίας. Γι' αυτό θέλουμε αυτές τις 50 δεσμευτικές ανώτατες τιμές. Και είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε σε αυτές τις ε, καρκινογόνες προτεραιότητες, να τις πούμε έτσι, αυτές που είναι σημαντικές για τις γυναίκες εργαζομένους. Το θέμα του φύλου είναι πολύ σημαντικό γενικότερα. Διότι η επαγγελματική καρκίνη για τις γυναίκες είναι αόρατη. Γιατί θέλουμε αυστηρότερες οριακές τιμές. Για ένα πολύ απλό λόγο. Εάν είναι εφικτό σε μια χώρα κάτι, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να, να γίνει εφικτό και αλλού. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Και κάτι άλλο. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογή και με τι αναπαραγωγικέ ε, τοξικέ ουσίε. Και διαφωνώ με την Κομισιόν επ' αυτού. Για πολλέ τέτοιε τόξο, όπω τι λέμε, ουσίε, δεν είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει κάποιο κατώτατο Για παράδειγμα, το μπιφενολ 2 ή ε, οι φθαλιούχε ουσίες. Όλες αυτές είναι επικίνδυνες ε, για την αναπαραγωγική διαδικασία και είναι και ενδοκρινικοί διαταράκτες, για, τις οποίους, για τους οποίους διαταράκτες δεν έχουμε ε, τιμή κατοφλίου. Άρα η συμπερίληψή τους εμέσως θα βελτίωνε την προστασία από αυτούς τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και υπενθυμίζω ότι οι ουσίες Reprotox ήδη συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής πολλών εθνικών μέτρων πρόληψης του καρκίνου. Και έχουμε και μία μελέτη επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δείχνει ότι υπήρξαν ωφέλη, για παράδειγμα στη Γαλλία και στη Γερμανία, από τη συμπερίληψή τους μεταξύ των εθνικών μέτρων κατά των καρκινογόνων ουσιών. Είναι σημαντικό λοιπόν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή και σε αυτές τις ε, τοξικές για την αναπαραγωγική διαδικασία ουσίες και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Ρεμπέκα Σμιθ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ξέρουμε ότι θα υπάρξει ένα πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύμα, άρα συνολικά είναι φιλόδοξη η πρόταση. Και υπάρχει ευρεία στήριξη και για την πρόταση και για τις ωραϊκές τιμές που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Και υπάρχουν και πολλές άλλες σημαντικές διατάξεις σε αυτήν την ε, οδηγία που θα ωφελήσουν τους εργαζόμενους. Στόχος αυτής της πρότασης και των επόμενων βημάτων είναι η καλύτερη προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνες στον τόπο εργασία, αλλά υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είπαν ορισμένοι πριν τον λόγο. Και είπαν ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό. Ως Business Europe είμαστε υπέρ νέων δεσμευτικών ορίων με του όρου που έθεσα προηγουμένως. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από την έκθεση σε αυτές τις ουσίες, όπως με οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα, αυτό είναι δυνατόν εάν είναι εφαρμόσιμο, αν οι εργοδότες μπορούν να την εφαρμόσουν. Και γι' αυτό είναι σημαντική η εφικτότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα τελευταία ομιλήτρια η Μαρίτα Ούλσκο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, ευχαριστώ για όλα τα στοιχεία και επιχειρήματα που μας δώσατε και όπως ε, είπα και στην αρχή είναι θέμα που μας ενδιαφέρει όχι μόνο ως πολιτικούς αλλά και ως ανθρώπινα όντα, γιατί όλοι έχουμε υποστεί τις συνέπειες ε, είτε στον εαυτό μας ή στο περιβάλλον μας του καρκίνου. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε όσο γίνεται την πρόταση της Επιτροπής. Μόλις ξεκινάει η διαδικασία αυτή και Θέλουμε να είμαστε αποφασιστικοί για να επιτύχουμε αποτελέσματα ευρείας κλίμακας που να έχουν επιπτώσεις στη ζωή και στην εργασία των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη. Φυσικά θα υπάρξουν αποκλήσεις, δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο αφετηρίας σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά Στόχος μας είναι να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη η πρόταση, η οδηγία. Και δεν θέλουμε μόνο κάποια πρωτοπόρα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με αυτή την οδηγία. Θέλουμε να γίνει κάτι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Δεν θα επιτευχθούν όλα ε, ευθύς εξ αρχής. Αλλά η οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίσει όσους θέλουν να κάνουν περισσότερα. Και φυσικά πρέπει να καλύπτει και τις γυναίκες και τους άνδρες εργαζομένους σε όλα τα τμήματα της αγοράς εργασίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και φυσικά θα είμαστε σε επαφή το επόμενο διάστημα ούτως ώστε να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μαρίτα. Θα ε, λοιπόν, 29 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε την έκθεση, 14 Δεκεμβρίου το μεσημέρι, τροπολογίες, 25-26 Ιανουαρίου θα μιλήσουμε για τις τροπολογίες, η ψηφοφορία θα γίνει 27-28 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συμμετασχόντες, τους ειδικούς. Η διαδικασία είναι πολύ σημαντική στις μελλοντικέ μας εργασίες και χρειαζόμαστε πάντα και τους ειδικού. Και προχωρούμε και πάμε στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης έσπιση του προγράμματος στήριξη διαφορετικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020. Ο εισηγητής έχει το λόγο, ο κύριος Τζάμπα Σόγκορο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ε, και τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες 300 περίπου που δείχνουν σαφέστατα τις ανησυχίες και το ενδιαφέρον για το έργο και τις απόψεις μας σχετικά με το τι πρέπει να αφορά. Καταρχήν οι ανησυχίες. Ορισμένες ε, τροπολογίες ε, έδειξαν κάποια επιφυλακτικότητα απέναντι στο πρόγραμμα ως εργαλείο για να επιβάλλει από πάνω πολιτικές στα κράτη-μέλη. Δεν πιστεύω όμως ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω, εις ό,τι αφορά την πολιτική, δεν υπάρχει τίποτε το κενό φανές, ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις βάσει συνθήκων των κρατών μελών ε, τους κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας ή τους κανόνες ε, για τις ε, εθνικές οικονομικές πολιτικές υπό την ευρεία καθοδήγηση του Συμβουλίου για να συμβάλλουν στους στόχους. Οι στόχοι του προγράμματος δεν αντιβαίνουν προς αυτό που οφείλει η χώρα στους πολίτες σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον για ανάπτυξη και απασχόληση ε, παροχή, ύπαρξη διακυβέρνησης, ε, διοίκηση, σωστή υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία κτλ. Υπ' αυτή την έννοια το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόσθετο εργαλείο στην εργαλειοθήκη μας για να πετύχει αυτούς τους στόχους και εξαρτάται από τα κράτη-μέλη αν θα το χρησιμοποιήσουν ή όχι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Πιστεύω ότι με τις, μέσω των τροπολογιών θα διασφαλίσουμε το νέο μέσο, θα διασφαλίσει μεγαλύτερο η αίσθηση ιδιοκτησίας από τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκομένους, θα γίνει διαφανέστερο και θα αντιμετωπίσει περισσότερα κοινωνικά προβλήματα. Ελπίζω ότι αν εγκριθεί το μέσο αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις όχι αφού υπάρξει κρίση, αλλά για την πρόληψη της κρίσης ώστε τα μέτρα που θα ληφθούν να μην οδηγήσουν σε ταλαιπωρία τους ευάλωτους. Ε, τώρα, για την ιδιοκτησία, τα κυβερνήσει των κρατών μελών θα πρέπει να αναλάβουν πλήρη ευθύνη των πράξεών τους. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να διατηρήσουν πλήρη ιδιοκτησία, να νιώσουν ότι είναι δική τους υπόθεση οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται και που έχουν συμφωνηθεί. Ε, να υπάρξει συνέπεια μέχρι την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Πολλές τροπολογίες πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση και το χάρηκα πολύ. Και συμφωνούμε ότι στη διαδικασία του καθορισμού των προτεραιοτήτων τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα είναι ίση, ισότιμη εταίρη για να υπάρξει μια συμφωνία που θα εγκριθεί και από τα δύο μέρη. Επίσης χαίρομαι γιατί σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες ε, προσέθεσαν ε, ένα στοιχείο στην ιδιοκτησία. Ε, μίλησαν για τις διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους για τις μεταρρυθμίσεις. Συμφωνώ ότι όταν αξιολογούμε το αίτημα για τεχνική βοήθεια, η Κομισιόν πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαδικασία διαβουλεύσεων που προϋπήρξε. Δεν πιστεύω όμως ότι πρέπει να πάμε τόσο μακριά ώστε να εφαρμόσουμε το, τους κανόνες των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων ε, που είναι περίπλοκοι κανόνες για περίπλοκες συμφωνίες εταιρικών σχέσεων και επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση ε, που διαρκεί και προγράμματα που διαρκούν ε, δεκαετίες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εδώ τόσο αυστηρέ οι προϋποθέσεις. Τώρα για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Χαιρετίζω ένα μεγάλο αριθμό ε, ε, τροπολογιών για το θέμα αυτό τις αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας που χρειάζονται οπωσδήποτε για την καλή λειτουργία του προγράμματος. Όμω, εν προκειμένου νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή ισορροπία. Για παράδειγμα, ακόμα και μέσα στα διαρθρωτικά ταμεία που ασχολούνται με έργα που είναι πολύ μεγαλύτερα, οι, ενημέρω... οι κανόνες για την ενημέρωση και τη δημοσιότητα ζητούν από τα κράτη-μέλη να δίνουν μια σύνοψη του έργου, ε, αρχή, τέλος και χρηματοδότηση και τόπο ε, ή ο στόχος του Ταμείου. Πολλές τροπολογίες και δικές μου έγιναν για την ενίσχυση της κοινωνικής πτυχής του προγράμματος, ενίσχυση της ε, πάλης κατά της ανεργίας, προώθηση της ε, κοινωνικής ενσωμάτωσης, εκπαίδευση καλή. Τώρα, για τους δικαιούχους, πολλές τροπολογίες επιμένουν ότι οι αρμόδιες αρχές ε, θα ε, πρέπει να ε, αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά. Οι μεταρρυθμίσεις Τώρα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ε, έχουμε επιμερισμένη ευθύνη. Ε, αυτό δεν πρέπει να το πειράξουμε. Ε, ένα θέμα είναι η φορολόγηση που είναι η κυριαρχία των κρατών μελών. Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό από την άποψη των στόχων του προγράμματος. Υπήρχαν και τροπολογίες που ζήτησαν το έργο να συμπεριλάβει φοροποφυγή, φοροδιαφυγή κλπ. Ε, υπήρξαν και άλλες τροπολογίες ε, ότι η πηγή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα να μην είναι προηγούμενο για το μέλλον, να μην συνιστά προηγούμενο. Θεωρώ ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση η Κομισιόν πρέπει να αναλύσει και την καταλληλότητα εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου προγράμματος για την περίοδο μετά το 2020. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα η εναλλακτική για τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στο χρηματοδοτικό φάκελο του προγράμματος με πρόσθετους πόρους. Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους για αυτό το πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα ήταν χρησιμότερο αυτή η εναλλακτική να παραμείνει ανοιχτή εδώ. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος ε, να υπάρξει συμβιβαστική λύση. Ναι, θα πούμε ή όχι σε αυτή τη δυνατότητα. Αυτά ήταν τα βασικά που ήθελα να πω σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους για τη συμβολή τους και θα περιμένω και άλλες απόψεις σας. Ελπίζω να μπορέσουμε να καλύψουμε ε, στις επόμενες συζητήσεις μας ε, πολύ, πολλά, όσο γίνεται περισσότερα θέματα. Ευχαριστώ. Σέρχιο Γκουτιέρεθ Πρέτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εργασία του και την καλή του θέληση για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ε, καταρχήν, ε, φυσικά συμφωνούμε με ένα πρόγραμμα βοήθειας προς τα κράτη-μέλη, για να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα πολιτικό θέμα και ένα θέμα χρηματοδότησης που είναι εντελώς διαφορετικά και πρέπει να επιληθούν με διαφορετικές μεθόδους. Το πιο σημαντικό από την πλευρά μου είναι το πολιτικό πρόβλημα, διότι σε τελευταία ανάλυση όλα συνδέονται. Ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για να εφαρμοστούν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις από ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ε, και του πολιτικού κόσμου τίθεται σε θέμα της ε, πολιτικής νομιμοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης που εισήχθη τα τελευταία χρόνια μέσω του 2 και του 6 Πρέπει δηλαδή να συνδυάσουμε το πρόγραμμα αυτό, να τεθεί και να εφαρμοστεί με βάση τις κοινωνικές ευαισθησίες που ε, συνδέονται με τα μέτρα αυτά που εισήχθησαν. Γι' αυτό κάναμε τροπολογίε για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ενημέρωση τη κοινή γνώμη, για να είναι γνωστό ποιοι είναι οι σύμβουλοι, ποιοι είναι οι τεχνικοί, ποιε είναι οι εταιρείε που αναλαμβάνουν να χορηγήσουν αυτή τη βοήθεια, να υπάρχει δημοκρατικό έλεγχο σε, σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό και τοπικό επίπεδο, να υπάρχει συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, γιατί σε τελευταία ανάλυση η τεχνική αυτή βοήθεια που πρέπει, όπως είπα, να ενταχθεί εντός των προγραμμάτων οικονομικής διακυβέρνησης που προωθείται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή μέσω των άλλων μέτρων που προβλέπει το 2-pack και το 6-pack. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν για να μην υπάρξει περισσότερη αναταραχή στην κοινωνία στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας και στο πώς την αντιλαμβάνονται γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν επιβληθεί. Και όπως σας είπα, πολλές φορές επιβλήθηκαν από τους νέους μηχανισμούς λόγω της οικονομικής κρίσης. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η πρόταση αυτή για να συμπεριλάβει αυτά τα στοιχεία που θα δώσουν περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση που σχετίζεται με την ε, αποδοχή από τους πολίτες και την διαφάνεια. Για αυτό σας τα εξηγώ όλα αυτά τα πολιτικά προβλήματα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για να διορθώσουμε σφάλματα του παρελθόντος και να προλάβουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Βεβαίω κύριε Ισηγητά, έχετε δίκιο. Οι μηχανισμοί αυτοί ήδη υπάρχουν και λειτουργούν. Για τα διαδοτικά ταμεία για παράδειγμα. Οπότε σε πολλά κράτη-μέλη για παράδειγμα να ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε ορισμένες χώρες αυτή η βοήθεια δίνεται κάπως ε, με τρόπο άτυπο. Είναι μια γκρίζα ζώνη. Πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι πρέπει να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση, λήψη υπόψη των ανησυχιών της κοινωνίας για να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Και δεύτερον, η χρηματοδότηση. Βεβαίως. Συμφωνούμε ότι είναι περιορισμένη η χρηματοδότηση στα πλαίσια του ευρύτερου ενωσιακού προϋπολογισμού. Αλλά αυτή η πρικοδότηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι γίνεται σε ένα ευαίσθητο πλαίσιο. Γιατί έχει να κάνει με τα δεθωτικά ταμεία που σχετίζονται με την αναδιανομή και την πολιτική συνοχής. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες και θέλω να προσέξετε τις τροπολογίες 144 και 145. Πρέπει να τίθονται όρια στις χρηματοδοτήσεις που μπορεί να κάνει τεχνική βοήθεια. Αυτό να μην αποβεί σε βάρος, για παράδειγμα, των χρηματοδοτήσεων του κοινωνικού ταμείου. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν με τον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή τώρα να αφαιρεθούν χρηματοδοτήσεις από κάποιο άλλο κράτος μέλος για να βοηθήσουμε κάποιο άλλο κράτος μέλος να εφαρμόσει τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, κάτι τέτοιο φαίνεται δυνατό όπως είναι τώρα η πρόταση και αυτό πρέπει να ε, περιοριστεί. Οπότε, ως σοσιαλιστική ομάδα θα κάνουμε τις προτάσεις μας για να επιτύχουμε μια συνένεση αλλά επειδή υπάρχουν πολιτικές ευαισθησίες πρέπει να υπάρχουν ρήτρε διαφύλαξης, πρέπει λοιπόν να περιοριστούν και να επανεξεταστούν και οι πιστώσεις πώς θα χορηγούνται. Αλλά συμφωνούμε ότι εάν υπάρξουν ε, επαρκείς προφυλάξεις, εάν υπάρχει επαρκής ε, σοφροσύνη, τότε Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και την τοπική αυτοδιοίκηση να εφαρμόσουν τι καλύτερε, επαναλαμβάνω, μεταρρυθμίσει, όχι αυτέ τι ιδεολειπτικέ που ορισμένοι θέλουν να μα επιβάλλουν. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαριάν Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή Είναι πολύ θετικό το σχέδιο πρότασης. Συμφωνώ με την προοπτική του σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα όταν μιλάει για την ανάγκη ε, θέσπισης προτεραιοτήτων για την απασχόληση και την παραγωγικότητα, ιδιαίτερα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Συμφωνώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να στοχεύσουμε για ένα ε, ευεπίφορο περιβάλλον ώστε να ωφεληθούν τα κράτη-μέλη από την πολιτική συνοχής και να βελτιωθεί και το ποσοστό απορρόφηση των κονδυλίων. Μία ερώτηση, γιατί αλλάξατε από 100% επιλέξιμο κόστος σε προαιρετικό από... Γιατί το κάνατε προαιρετικό το όριο αυτό, το επιλέξιμο κόστος. Επίσης, κάποιοι συνάδελφοι έχουν ανησυχίες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, ίσως στα πλαίσια της τάσης της Κομισιόν. Είναι ευαίσθητο για την πολιτικό το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό το τελικό μας έγγραφο να διευκρινίζει ότι πρόκειται για εταιρική σχέση που καθοδηγείται από τα κράτη-μέλη και λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες των πολιτών και πρέπει να διασφαλίσουμε την διαφάνεια και το, την ε, προσπάθεια ε, να εφαρμόσουν το πρόγραμμα ε, κοινωνική συμμετοχή δηλαδή. Μου φαίνεται ότι μπορούμε να βρούμε ένα χώρο, ένα κοινό έδαφο, έδαφος εδώ. Τα σχόλια του εισηγητή για την ιδιοκτησία, για το να νιώσουν ότι είναι δικά τους, είναι πολύ σημαντικά στη συνολική εικόνα και συμφωνώ να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση της στόχιας, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αναφέρατε και άλλα, και άλλους κοινωνικούς στόχους που θα πρέπει να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα. Δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να διεδώ προσεκτικά τις ε, συμβιβαστικέ τροπολογίες, αλλά με χαρά θα συνεργαστώ πάνω σε αυτά με τον εισηγήτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, εισηγητή που πρότεινε τροπολογία συμβιβασμού. Εγώ είμαι σκιώδης και για αυτή την έκθεση, για αυτό τον κανονισμό στην Επιτροπή Ρέτζη και είχαμε εκτενείς συζητήσεις γιατί είναι ένα πρόγραμμα που αφορά και τις ε, ομάδες τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα και την Κύπρο και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλες ε, χώρες. Η Ρέτζη μετέβη στην Ελλάδα λίγες εβδομάδες πριν και αυτοί που εργάζονται επιτοπίως, δηλαδή που εφαρμόζουν το πρόγραμμα στην Ελλάδα, και όταν δούμε και την έκθεση του ελεγκτικού δικαστηρίου, βλέπουμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι επιτυχές για την εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής, αλλά υπάρχουν λήψεις και κενά σε, άλλες, σε άλλους τομείς και πολιτικές. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό μέσο για τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη την ε, πραγματική και σωστή εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων. Και η ομάδα μου θα υποβάλει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν ε, μιλάμε για την πραγματική χρήση αυτού του μέσου γιατί στις χώρες ε, υποπρόγραμμα είδαμε ότι υπήρχε θέμα λογοδοσίας από οργανισμούς που δεν είχαν ενταχθεί σαφώς ε, σε αυτό το πλαίσιο. ως προς την δημοκρατική νομιμότητα και τη λογοδοσία. Και βεβαίως αυτό σχετίζεται και με τον κώδικα δεοντολογίας και την αρχή της εταιρικότητας. Ίσως σας παρανόησα, ε, κυρία Ισηγητά, γιατί εδώ μιλάμε για κανόνες όπου συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει μια συμμετοχική διαδικασία λοιπόν και είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να τονιστεί περισσότερο στις τροπολογίες συμβιβασμού. Το θέμα της ε, κοινωνικής συμμετοχής, την έλλειψη αποκλεισμών και την ε, συμμετοχή των τοπικών αρχών, επίσης το συζητήσαμε και μπορούμε να αποστείλουμε έτσι ένα μήνυμα και προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έτσι ώστε αυτό το μέσο να χρησιμοποιηθεί στα κράτη-μέλη, από τα κράτη-μέλη, όπως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Dominique Martin. Κατανοείτε ότι δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας και ο αριθμός των τροπολογιών μου δείχνει ότι πολλοί συμμερίζονται την άποψή μου. Αυτή η τεχνική αρρωγή μετά από αίτημα των κρατών μελών ε, για τα προγράμματα στήριξης και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται κάτι το καλό, συμπαθητικό. Γιατί όχι. Αλλά νομίζω ότι αποτελεί ένα μέσο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν εθνικές αρμοδιότητες, όπως την εκπαίδευση, την ε, πολιτική, ε, την γενικότερη εθνική πολιτική και το θέμα των μεταναστών. Δηλαδή δίνουμε επιπρόσθετα προνόμια σε ορισμένες κατηγορίες και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προβεί σε συστάσεις που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν και γιατί θα πρέπει να τις εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Για να τους, δοθούν, να τους δοθεί ειδική οικονομική ε, βοήθεια. Δηλαδή, στην ουσία τους κρατάει στο χέρι η Επιτροπή. Αυτό το παιχνίδι παίζεται. Κάτι το οποίο είναι εντελώς τρευλωτικό. Ευχαριστώ. Οπότε, Νομίζω ότι δεν ε, θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ποιος θέλει να πάρει το λόγο και με ενοχλεί το ότι έχω πολλά ονόματα. Ε, με συγχωρείτε, περίμενα να καταλάβω λίγο Βιτσέντσο Μπακάρο. Είμαι από την υπηρεσία που ασχολείται με αυτή την υπηρεσία. Είμαι νομικός σύμβουλος της υπηρεσίας αυτής. Ευχαριστώ όλους τους ε, αξιότιμους βουλευτέ για τη συζήτηση και τις τροπολογίες που υπέβαλαν και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που ανέφερε και εκείνος. γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα εξ αυτών. Το πρόγραμμα αυτό εκτελείται μόνο μετά από αίτημα του κράτους μέλους. Μόνο αν μας υποβληθεί αίτημα χορηγείται αυτή η βοήθεια. Και το αίτημα αυτό για στήριξη σε ορισμένου τομείς που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση ή με μεταρρυθμίσεις που θέλουν να εφαρμόσουν με την πρωτοβουλία τους των κρατών μελών. Μετά το αίτημα υπάρχει διάλογος μεταξύ του Κοινοβουλίου και, ε, συγγνώμη, της Επιτροπής και του κράτους μέλους για να καθοριστούν προτεραιότητες, για τα μέτρα στήριξης και τη χρηματοδότηση που χρειάζεται η εφαρμογή αυτών των μέτρων στήριξης. Επίσης να διευκρινίσουμε ότι η χρηματοδότηση για, την, ε, για τα μέτρα αυτά δεν είναι κάτι που χορηγείται στα κράτη-μέλη, δεν είναι χρηματοδότηση προς το κράτος μέλος, είναι μια χρηματοδότηση για να πληρώσουμε τους εμπειρογνώμονες που θα αξιοποιηθούν στα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν το κράτος μέλος να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό για τον τρόπο χρηματοδότησης. Αν δηλαδή αφαιρούνται αυτές οι χρηματοδοτήσεις από τις εθνικές χρηματοδοτήσεις, από τις χρηματοδοτήσεις προς τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων για παράδειγμα. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Για, τώρα για τους στόχους του προγράμματος. Όπως αναφέρει η γνωμοδότηση του κυρίου Σόγκορ και άλλες τροπολογίες, στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει την εφαρμογή πολιτικών που έχουν εγκριθεί μέσω άλλων νομοθετημάτων της Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι ε, μια νέα πολιτική, βοηθάει την εφαρμογή άλλων πολιτικών. Άρα πρέπει να υπάρχει αποδοχή από πλευράς του κράτους μέλους, όπως υπόθηκε σαφώς. Και η αποδοχή προκύπτει από το ότι το ίδιο κράτος μέλος κάνει το αίτημα. Μετά γίνεται διάλογος με την Επιτροπή. Και όταν το κράτος μέλος διατυπώνει το αίτημα, κατά πάσα πιθανότητα έχει κάνει διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο με όλους τους ενδιαφορομένους ε, και σε εθνικό επίπεδο και φυσικά και κατά πάσα πιθανότητα διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών. Τώρα εμείς ως κράτος μέλος δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν έχει γίνει αυτή η διαβούλευση. Γιατί αυτό είναι θέμα ε, αρμοδιότητας του κράτους μέλους και τα κράτη-μέλη έχουν ε, τη δική τους ε, νομιτάξη, τις διαδικασίες τους. Η Κομισιόν δεν μπορεί να δράσει ούλτρα να υπερβεί τις, δραστηριότητες, τις αρμοδιότητες της, οι οποίες περιορίζονται στη συζήτηση με το κράτος μέλος για το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. Άρα το θέμα της αποδοχής από τη χώρα είναι βασικό. Κάτι άλλο. Διαφάνεια λογοδοσία. Βεβαίως ε, θα ενεργήσουμε με πλήρη διαφάνεια έναντι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ήδη στην πρόταση περιλαμβάνεται η υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει στο τέλος κάθε χρόνου για να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας έναντι των άλλων θεσμικών οργάνων από τη μία και από την άλλη μεριά ε, λόγω του περιορισμού του προγράμματος, του, των περιορισμένων διαστάσεων. Ευχαριστώ πολύ, αλλά αν έχετε άλλες ερωτήσεις ε, να επανέλθω. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ίσως ό,τι αφορά την νήξη ότι η Κομισιόν θέλει να ανακατευτεί στα κράτη-μέλη και στις υποθέσεις τους. Ευχαριστώ θερμά την Κομισιόν για τη δήλωσή της. Ε, μία ερώτηση. Ε, είπατε ότι κατά την παρακολούθηση των ε, του τρόπου δαπανών των ε, κονδυλίων της Ένωσης. Δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα, έτσι είπατε. Και μιλήσατε και για τις κοινωνικές διαβουλεύσεις. Ότι αυτές δηλαδή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, στις διαβουλεύσεις και στη χρήση ενωσιακών κονδυλίων πρέπει να φροντίσουμε ότι θα γίνονται διαβουλεύσεις σε κάθε κράτος μέλος ε, γιατί ζούμε σε περίοδο μάλλον βαθιάς κρίσης και οι πολίτες δεν έχουν πολύ εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι όταν γίνονται διαβουλεύσεις για τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τι μέσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες, η κοινωνία μέσα της Ένωσης, αυτά πρέπει να γίνονται γνωστά, χρειάζονται διαβουλεύσεις. Και Ρωτώ την Κομισιόν. Δεν πρέπει τα κριτήρια για τη χρησιμοποίηση κονδυλίων να συμπεριλαμβάνουν και την υποχρέωση διαβουλεύσεων στα κράτη-μέλη. Ε, ο εισηγητής και πάλι, ο κύριος ε, Σόγκορ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ε, επαναλαμβάνω, συμφωνώ με την λογοδεσία με την Κομισιόν, δεν θα τα επαναλάβω. Εμείς θα περιμένουμε να γίνουν και οι επόμενες συζητήσεις και για την ερώτηση της κυρίας Χάρκιν. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνέπεια με την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ψηφίσουμε στις 8 Νοεμβρίου στην ΕΜΠΛ. Στη Ρέγγι θα ψηφίσουν στις 29 Νοεμβρίου. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης, τα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Ε, οι επόμενες συνεδριάσεις στις 7 Νοεμβρίου 3 με 6.30 το βράδυ και 8 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι το 12.30 και 3 με 6.30. Ε, καλή σας ημέρα, σας χαιρετώ. Καλές εργασίες.